Delange, she's not here. I don't know. I'm waiting for Esther. Περιμένουμε την Esther. Για το βασικό σημείο της Έστερ Delange πρέπει να έρθει. We have just three socialists. call her. We will vote anyway. Okay. Um, io penso che possiamo Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημείο 5 της ημερής τετάξης Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφού ψηφίσαμε στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας της 3ης Σεπτεμβρίου τις τροπολογίες μας Όσον αφορά τις γραμμές του προπολογισμού, γραμμές του, συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού, σημερινή μας ε, αρμοδιότητα καθήκον είναι να εγκρίνουμε την γνωμοδότηση που συνοδεύει τις τροπολογίες. Έχουμε 20 τροπολογίες όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης που συνέταξε συνάδελφος Έστερ Ντελάνγκε, η οποία καταφθάνει. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Αν έχετε όλοι την κάρτα για τις ψηφοφορίες την κάρτα σας. Δεν έχετε κάρτα. τάσω στις χειρός θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε τότε. Ehm, Ψηφίζουμε με το χέρι. τάσω στις χειρός. Πώς το λέμε σπανικά, σαν τα δαμάνω μάνα. Λοιπόν, όλοι έτοιμοι. Ξεκινάμε στη ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Ποιος είναι υπέρ της 5. Κατά. Θα κάνουμε παλήθευση. Χρειάζεται παλήθευση. Ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος. Un Πέρας. Δεν το... Πρόεδρε. Η διερμηνία λέει ότι παράγραφος Πέντε μα είπε. Όχι, τροπολογία λέει ο πρόεδρο. Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώ τι ψηφίζουμε. Τροπολογία 5 λέει ο πρόεδρο. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 με το χέρι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 Γιέγκλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κύριε Ρόντοστ για την τροπολογία 17 υπάρχει η λέξη απελευθέρωση εγώ θα ήθελα αντί για απελευθέρωση να μιλάμε για ρύθμιση. Αν γίνει αυτό, τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία. Ρύθμιση αντί για απελευθέρωση. Ευχαριστώ, Ουλρικέ. Θα έλεγα ναι, διότι η Ελέζα έγνευσε θετικά. Δέχεται αυτή τη διόρθωση. Τροπολογία 17 μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Είσαι αντίθετος με τη διόρθωση. Ο κανονισμός λέει ότι αν κάποιος είναι αντίθετος με αυτή την τροποποίηση την προφορική δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ε, η Ελίζα ζητά το λόγο. Ich, ε, verstehe, du ε, Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Νίκολσον. Μετά από μια συζήτηση με την Ουλουρική και Ρόντους και τους σοσιαλιστές, εγώ συμφωνώ ότι στα γαλλικά υπάρχει μια γλωσσική δυσκολία. Μόνο στα γαλλικά είναι αυτό το πρόβλημα. Και μπορούμε ίσως να βρούμε μια άλλη διατύπωση για να λύσουμε το πρόβλημα στα γαλλικά. Σε επίπεδο ουσίας έχουμε ακριβώς την ίδια θέση. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας. Ε, George, οι φιλελεύθεροι συμφωνούν με αυτή τη διευκρίνηση της Ελίζαμπεθ ή εξακολουθείτε να είστε αντίθετοι όσον αφορά με τροποποίηση του κειμένου. Ε, ε, ε, φιλανθρωπήσει και να γίνει ρύθμιση είναι αντίθετες οι έννοιε στα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αυτή την αλλαγή. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Αλίμονο. Ούλρικα. Δεν είναι πρόβλημα ουσία, είναι ένα πρόβλημα καθαρά γλωσσικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη management, διαχείριση για το γερμανικό κείμενο σας λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να υποστηρίξω αυτή την τροπολογία. Στα γαλλικά όμως είναι αμφίσιμο. Αν μιλήσουμε για διαχείριση, management, νομίζω ότι όλοι μπορούν να το αποδεχτούν. Uh, Περιμένουμε ακόμα την άποψη των φιλελευθέρων. Αν δέχονται ή όχι διαφορετικά δεν μπορούμε να Άγνιο. έχοντας μητρική γλώσσα τα αγγλικά, η λέξη απελευθέρωση, διαχείριση και ρύθμιση όλα σημαίνουν πολύ διαφορετικά πράγματα και δεν μπορούν να ανταλλαγούν, να χρησιμοποιηθούν η μία έννοια αντί τη άλλη στη γλώσσα μα. Εντάξει, σαφέ λέει ο πρόεδρο, Εν αυτή αυτή περιπτώση, σύμφωνα τον κανονισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία τροποποίηση. Θα πρέπει δυστυχώ αλλήμω να τροποποιήσουμε την τροποποίηση 17 να την ψηφίσουμε όπω προτάθη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 17 άνευ τροποποίησεω. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 18. Υπέρ. 18. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο το τροποποιημένο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια στην Έστερ και σε απουσιάζει περνάμε τώρα στο σημείο το επόμενο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης ενδιάμεση έκθεση όσον αφορά τη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Λοιπόν, συνάδελφοι, άλλαξα κάπως το κείμενο της νομοδοτήσεως, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις θέσεις που επανειλημμένα εξεφράστησαν στην Επιτροπή μας, ενιαία, δηλαδή να ζητήσουμε στη γνωμοδότηση κόμμα κόμμα-αγκρή... να ζητήσουμε ένα πάγωμα του προϋπολογισμού της ΚΑΠ ε, σε πραγματικούς όρους ε, διότι η πρόταση Λεβαντόφσκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί περικοπή όμως ε, και όχι πάγωμα. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τη συζήτηση 3 Σεπτεμβρίου όπου εκεί έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις συναδέλφων όπως τον George Lyon, Esther DeLange κλπ. Ήθελα να προσθέσω την τροπολογία 18 τροπολογία 18 που προτείνει στην περίπτωση και άλλων περιποκών του ευρωπαϊκού προπολογισμού προϋπολογισμός για την κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούστε με ένα λεπτάκι. Τώρα, κάποιοι συνάδελφοι παρουσίασαν και την τροπολογία 16, η οποία δέχεται ουσιαστικά σαν βάση διαπραγματευτική την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό διότι και είναι η μοναδική τροπολογία επί της οποίας ίσως να υπάρξει κάποια, κάποιος προβληματισμός. Είναι σημαντικό επ' αυτού του σημείου όσον αφορά την τροπολογία 16 η Επιτροπή μας να ψηφίσει και να τοποθετηθεί με σαφή τρόπο ε, εν ώψη των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εκείνο που είναι υπέρ τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προτάσεις Λεβαντόφσκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προπολογισμό της ΚΑΠ θα πρέπει να υπερψηφίσει την τροπολογία 16. Για όλους εκείνους θέλουν αντιθέτως να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ζητώντα πάγωμα σε πραγματικούς όρους να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός θα πρέπει να καταψηφίσουν. Συγγνώμη που ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση και πάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Ο Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ένα σχόλιο έχω κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται περί του προϋπολογισμού. Μιλάμε εδώ για μείωση, περικοπές έτσι, του προϋπολογισμού. Διότι υπάρχουν αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι των νέων κρατών μελών και έχουμε και μελλοντικέ διευρύνσεις. Λοιπόν και οι γεωργοί, κυρίως των 15 παλαιών κρατών μελών, δέχονται πληροφορίε από τι οποίε αυξάνεται ο προπολογισμό, ενώ στην πράξη μειώνεται ο προπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι εδώ πρόκειται περί περικοπή μειώσεω του προπολογισμού. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο, είναι όλα ξεκάθαρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, ακόμα μια φορά, διανατάσσεω τη χειρό, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 λαβία και άλλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία Τροπολογία 8 απορρίπτεται. Κάνουμε έλεγχο. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Ξανά την 8. Τροπολογία 8 επαλήθευση. Έλεγχος. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 8. Υπέρ. Κατά. Άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Σεγγερία και υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία είναι μεγάλη διαφορά λέει ο πρόεδρος από αυτή τη γωνία βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ψήφοι διαφορά τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεν φαίνεται έλεγχος έλεγχος για τη 12 παρακαλώ ποιος είναι υπέρ της 12 Hausling υπέρ Αθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο. Ξεκινάει ψηφοφορία για την τροπολογία 12, ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη 12. Ψηφίσατε όλοι. Καλώς. Τέλος Τροπολογία 12 εγκρίνεται. Έχετε δίκιο. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος για τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Ξεκινάει ψηφοφορία, ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Στην 15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Προσοχή για τη 16, όπω σα υπενθύμησα. Ποιο ψηφίζει υπέρ θέλει διαπραγματευτική βάση να είναι αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όποιο ψηφίζει κατά προτιμά αυτό που είπε ο κ. Σεγκερέσκη ένα πάγωμα σε πραγματικού όρου. Δηλαδή να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμό. Τροπολογία 16 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Ποιο απέχει, είναι πρόεδρο, ποιο είναι κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Η 19 ε, καταπέφτει. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά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 Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 27 σε Κεριέσκη. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τέλος τροπολογία 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία του κειμένου σε τροποποίηθη. Όλοι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Πάει και αυτό. Πάντα υπάρχει κάποιος αντίθετος. Μισό λεπτό. Πρέπει να μετρήσουμε ακριβώς τον αριθμό των ψηφισάντων και πώς ψηφίσαν τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία της νομοδοτήσεως που τροποποιήθηκε. Ποιος είναι υπέρ. Σηκώστε τα χέρια και κρατήστε τα πάνω τα χέρια για λίγο. Μερικά δευτερόλεπτα. Κατά. Η πράσινη είναι κατά. Τέσσερις ψήφοι κατά. Αποχές υπάρχουν. Υπάρχουν αποχές. Όχι, όχι Τζιμ. Τρεις απόχες. Ωραία. Να έχετε ενία θέση παρακαλώ στην, στην αίθουσα. Sorry. Andiamo al punto 7 all'ordine. Σημείο 7 της ημερήσια διάταξη, τροποποίηση του κανονισμού 3 του 2008 του Συμβουλίου σχετικά με νέες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες. Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Μποβέ. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοδοτήσεως. Ο Χωσέ έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Just, uh, uh Θέλω να πω δύο λόγια πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε βέβαια την γεύση στην Ευρώπη. Σχετικά με το κείμενο αυτό τώρα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, θέλουμε να προωθήσουμε τρόφιμα ποιότητας, ανάλογα από πού προέρχονται και όχι με μια γενική παραγωγή, την βιώσιμη παραγωγή επίσης και θέλουμε να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην παραγωγή και τον πολίτη. Έπειτα, η οριζόντια διάσταση να μην οδηγεί σε διατροφικές κρίσεις. Τροπολογίες κατατέθηκαν πολλές, συχνά για τις αγορές τρίτων χωρών, για να πούνε ότι πρέπει να προωθείται και αγορά τρίτων χωρών. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα. 2007 με 2010 για παράδειγμα υπάρχουν προγράμματα για τις εξωτερικές αγορές που ήταν το 29% και 26% σε πραγματικά νούμερα για την προώθηση τέτοιων προγραμμάτων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε διάκριση. Ο στόχος δεν είναι μέσα από αυτό το κείμενο και να διαχειριστούμε την εσωτερική διάσταση αλλά και την εξωτερική, αλλά να προωθήσουμε τοπικά προϊόντα σε σχέση με την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και εγώ υπέβαλα τις δικές μου προτάσεις ως εισηγητής, οπότε εφόσον συμφωνείτε έτσι πρέπει και να ψηφίσετε και ανάλογη είναι και η στάση μου απέναντι στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Αυτά για να σας εξηγήσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύω. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι εγώ θα δεχτώ ότι αποφασίσει το σώμα. Καλώς ευχαριστώ, Χωσέ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ας προχωρήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες σήμερα. Διανατάσεις χειρός πάντα. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές ένας έλεγχος παρακαλώ. ηλεκτρονικός έλεγχος η τροπολογία 10 λαβία υπέρ. Συγγνώμη, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. Είχατε δίκιο. Τροπολογία 11. Παπαστάμκος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ντάντσιλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, περιμένετε. Τροπολογία 16. Υπέρ. Τροπολογία 16 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ε... Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται απορρίπτεται τροπολογία 3 απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 20 κότα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που τροποποιήθηκε υπέρ κατά κατά κατά αποχές δύο ψήφοι κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα υπέρ κατά Κρατήστε ψηλά το χέρι. Κατά. Μία ψήφος. Αποχές. Εσύ Λουίς απέχεις. Όχι. Ψήφος υπέρ. Και τελική ψηφοφορία για την έξοδο διαπραγματεύσεων υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλώς. Ευχαριστώ. Και η έκθεση Μπόβε ενεκριθεί. Συνεχίζουμε με τις εκθέσεις. Πάμε στο σημείο 8. Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την πρόθεσή τους. Μια στρατηγική για την πρόθεση των γεύσεων της Ευρώπης. Αφού έγινε ανταλλαγή απόψε όσον αφορά το θέμα, ε, ε πρέπει να ψηφίσουμε από την πρόταση πρωτοβουλία. 105 τροπολογίε είχαμε. Θα επανέλθουμε στην προβληματική και περιμένουμε και άλλες νομοθετικές ε, προτάσεις. Ζωζέ, θες ε, να, να προσθέσεις κάτι? Ωραία, τέλεια. Ξεκινάμε ψηφοφορία πάντα διανατάσσω της χειρός. Τροπολογία 35. Πατράω Νέβες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. 36. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 όχι 37 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 37 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με ανάταση χειρών. 38 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Όχι. Έχει εκπέσει. Συγγνώμη. Πέφτει και η 40. Καταπίπτει 43. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 46 εκπίπτει 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην... Ε, πάμε στην 53 με ένα ελαφρό άλμα. Ψήφι υπέρ της 53. Κατά. Αποχές. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 Ναι, ναι.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 αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά απόχέ, α εδώ πέρα αλλάζουν τα πράγματα μια στιγμή 73 ποιος είναι υπέρ κατά πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 73 άρχεται η ψηφοφορία Άρχεται. Έληξε. Πράγματι με μία ψήφο έχει απορριφθεί. 18-19. Απερίφθη 73. 72 Γκάμπριελ. <clears throat> με ανάταση χειρών. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ Θέλετε έλεγχο στην 72. Πάμε. Ηλεκτρονικό έλεγχο στην 72. Άρχεται η ψηφοφορία. 72. Το ΕΛΚ έχει ένα παραπάνω που ψηφίζει από ό,τι επιτρέπεται. Περισσεύει ένας βουλευτής του ΕΛΚ στις ψηφοφορία, τώρα είναι εντάξει. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφία. Ο κύριος Άγνιου. Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι υπήρχε μια πρόσθετη ψηφοφορία ένα που ψηφίζει παραπάνω από το ΕΛΚ λόγω τη ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά όταν γίνεται διανάταση χειρών η ψηφοφορία, Πώ ξέρετε ότι δεν υπάρχει ένα πρόσθετο από το ΕΛΚ. Μα δεν είχαν ποτέ αμφιβολίες για το θέμα αυτό, γιατί ήταν μεγάλε οι διαφορέ. Όπου υπάρχει, ψηφο... υπάρχει ε, μικρή διαφορά, τότε κάνουμε έλεγχο. Η 72 λοιπόν απερίφθη, τώρα ψηφίζουμε την 74. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 76 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Όλοι και όλες. Πέρας. Εγκρίνεται, ωραία, ωραία. 78 με ανάταση χειρών. 78. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 εκπιπτή πάμε στην 80 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές μια στιγμή 81 υπέρ κατά καταρχήν εγκρίνεται γιατί το έχει προτείνει ένας αντιπρόεδρος αλλά χρειάζεται και ένας ηλεκτρονικός έλεγχο στην 81. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία 81 Παπαστάμκος. Ψήφισατε όλοι, όλες. Εντάξει, πέρας. Εγκρίνεται, ωραία. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 84, 85 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απολύτωται, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 88. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία ελέγχου στην 88. Εντάξει, ψηφίσαμε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90. Εκπίπτει. Πάμε στην 93. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικό έλεγχο παρόλα αυτά για την 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται, ωραία. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 95 και 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιο έλεγχο η ηλεκτρονικό έλεγχος για 95 και 96 Νίκολσον Πατράου Νέβες άρχιε ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 97 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 98 έχει εκπέσει. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογικές αναφορές 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 3. Η 4 υπέρ κατά α, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7, ε, όχι θα την πει 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 11. Η ηλεκτρονικά για την σκέψη υπαριθμών 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Όχι, όχι, έχει εκπέσει όπως και η 13. 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 εκπίπτει 20 υπέρ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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 εγκρίνεται 30 και 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία στην έκθεση όπω έχει τροποποιηθεί όλοι υπέρ κατά υπάρχει κάποιο κατά ναι ναι ωραία αποχές όχι Συγχαρητήρια στο Ζωζέ Μποβέρ. Και τώρα πάμε στο σημείο 9. Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δεστητήτων που σχετίζονται με, τις με τη χρήση της γης και την δασοκομεία. Η Τζούλι Γκέρλινγκ είναι η συγγήτρια που τη βλέπω παρούσα. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοδότηση τη Τζούλη επί τη προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προδιαγραφέ για του λογιστικού κανόνε και σχέδια δράση για τι εκπομπέ και τι απορροφήσει αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τι χρήσει γη. Έχουμε 29 τροπολογίε που προτάθηκαν από την κυρία Γκέρλινγκ και άλλε 50 τροπολογίε υπευλήθησαν από άλλου βουλευτέ. Αυτέ οι νέε τροπολογίε προτείνουν λογιστικοί κανόνες για τη διαχείριση των διαφόρων τόπων βοσκής. Δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά επιβάσει ε, εθελοντική. και ότι οι εκπομπέ και απορροφήσει που οφείλονται στην απορρόφηση υδάτων από τι υγρέ περιοχέ και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των κρατών μελών. Και εκπομπέ των αερίων θερμοκηπίων και θερμοκηπίου και από ανθρωπογενεί δραστηριότητε. Κάποιε τροπολογίε θετούν και ε, την κανονική διαδικασία έναντι κατοξεσδότηση πράξεων. Θες το λόγο, Τζούλη. Όχι, ψηφίζουμε. Ξεκινάμε, συνεχίζουμε να διανατάσσουμε στις Τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ. Α, συγγνώμη. 39. Τροπολογία 39, υπέρ. Κατά. Τροπολογία 39. Έλεγχος. Ηλεκτρονικό έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 39. Votato tutti. όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Όχι. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 44. Μαγκίνες Ντελάνς. ξεκίνα η ψηφοφορία. Ο έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Προσοχή με το ΕΛ και ότι υπάρχει ε, μία ψήφος παραπάνω. Με μεγάλη πλειοψηφία ανεκρίθη. 28-13. Τροπολογία 46 υπέρ. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48. 48 και 49. Έκουτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Αμισό λεπτό. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ κατά μισό λεπτό. Κατά. Ποιος είναι κατά της 15. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Τροπολογία 15. Ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 15 του συγητού. πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 17. 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 και 53 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 54 καλνιέται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 της ηγήτριας υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 58 υπέρ κατά μισό λεπτό έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 58. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Μαγκίνες Δελάνος. Υπέρ της 60. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια διαφορά. 23 υπέρ. Τις τροπολογίες 23 ηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 25 όχι ναι 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 τροπολογία 63 όχι Πάμε στην τροπολογία... Α, τις αφήνουμε όλες. Τροπολογία 30 πάμε. Υπέρ. Πάμε σε τελογικές σκέψεις. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Δεν αρκεί. Αγκρίνεται. Εντάξει. Τροπολογία 1 της γήτριας. Όχι, καταπίπτει. 31 της ηγήτριας. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 35. 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 36 όχι. απορρίπτω. Τροπολογία 2 πάμε. Υπέρ, κατά. Να κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 2. Ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινά. η τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Γιατί δύο. πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 37, όχι. Πάμε στο τέλος. Τελική ψηφοφορία στον αφορά το σχέδιο γνωμοδότης που τροποποιήθηκε. Ποιος είναι κατά. Κατά. Κατά. Μόνο κατά παρακαλώ. Αποχές. Αποχές παρακαλώ. Τέλεια. Πέρας. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έχουμε το σημείο 10 της σημερινής διάταξης. Τροποποίηση της απόφασης 2008-971 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του δασικού που πολλαπλασιαστικού υλικού της κατηγορίας χαρακτηρισμένου στο πεδίο εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και στην επικαιροποίηση του ονόματος των αρχών που είναι αρμόδιες για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής. Συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πολύ τεχνική φύσης το θέμα και απλουστευμένη διαδικασία που αποφασίσαμε ε, πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί να προχωρήσουμε γρήγορα εκτός αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που επιθυμεί να πάρει το λόγο για το σημείο 10? Όχι. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την απιστευμένη διαδικασία λοιπόν. Καλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Αναλόγως έχουμε το σημείο 11 τη ημερήσια διάταξη. Συζητούμε την παράταση περίοδου εφαρμογή που προβλέπει απόφαση 2003-17 του Συμβουλίου για επικαιροποίηση των ονομασιών της θήτης χώρας και των αρμοδίων για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής αρχών. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο εκθέσεων αφορά την πρώτη αποφάση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τέτοια απόφαση έδωσε έναν κατάλογο τρίτων χωρών για την εισαγωγή διαφόρων ειδών φυτών και για ε, σπόρων κλπ. Λοιπόν, η, η περίοδος κατά 10 χρόνια παρατείνεται. Μισό λεπτό να προσέξετε, θα προχωρήσουμε γρήγορα. Η θέση σε ισχύ τη νέα απόφαση θεωρείται ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη για να εγγυηθούμε την αναγκαία προμήθεια των διαφόρων σπόρων στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δυστυχώ όμω, συνάδελφοι, δεν, υπα... δεν είναι να εφαρμοστεί εδώ η προστευμένη διαδικασία όπω κάναμε και για το σημείο το προηγούμενο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σε τις παλαιές διατάξεις επιτροπολογίας με το σύστημα των κατεξοδότησης πράξεων και για την εκτέλεση των συνθήκων. Γι' αυτό το λόγο προτείνονται δύο τροπολογίες που αφορούν μόνο και αποκλειστικά την επιτροπολογία. Μετά από άλλες συζητήσεις και επαφές με την νομική υπηρεσία των τριών θεσμικών οργάνων, εντωμεταξύ έχω την πρόθεση να παρουσιάσω μια τροπολογία περισσότερο για λόγους νομικής τυπικότητας και μόνο ένα σημείο για να εξηγήσω του λόγου ε, για τι άλλε δύο τροπολογίε. Δηλαδή τα άθρα όσον αφορά την παλιά επιτροπολογία θα πρέπει να διαγραφούν διότι είναι ασύμβατα ε, με το σύστημα των αξιοσωτήσεων πράξεων και τις αρμοδιότητες εκτελεστικές που προβλέπονται από τις νέες συνθήκες της Αβώνας. Κατά λοιπά προτείνω να γίνει αποδεκτή η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την παρούσα μορφή δοθήση της σημασία του θέματος και του κατεπήγοντος χαρακτήρα. Δεχόμαστε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής αλλά πρέπει να τροποποιήσουμε αυτά τα δύο σημεία που αφορούν τι εφαρμοτικέ πράξει τη ε, Λισαβόνα που δεν έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν συμφωνείτε, θα προχωρήσουμε με ο τρόπο, εκτό αν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θέλει να πάρει το λόγο. Ουχή. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουν να πάρουν το λόγο, μήπως όχι. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 19 Σεπτεμβρίου, αύριο στις 12 το μεσημέρι. Δεν υπάρχουν ε, συνάφιους, ζήτησαν το λόγο. Λοιπόν, προθεσμία είναι αύριο για τυχόν τροπολογίες. Αν δεν υπάρχουν τροπολογίες θα προχωρήσουμε όπως αναφέρθηκε. Σημείο 12. Πάμε στο σημείο 12 της ημέρας διάταξης, δηλαδή στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες συζητήσαμε τον Τεν την ε, ΚΟΑ, την ΕΝΙΑ και συνεχίζουμε τις εργασίες με τη δεύτερη έκθεση του, του κ. Κάπουλα Σάντος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Υπενθυμίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση έχουμε πάνω από 2.000 τροπολογίες και, αν, και γίναν συζητήσεις επίμαχες επί του θέματος, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλές τροπολογίες που ακολουθούν παρόμοια κατεύθυνση. Ε, θα δώσω το λόγο παρευθύ στο συνάδελφο Λουίς Κάπουλα Σάντο. Χαιρετίζω και το διευθυντή Πλέμπακ της Γενικής Διευθύνσεω Γεωργίας που κατέφθασε. Και Λουίς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, πρόκειται για μία πρόταση κανονισμού, η οποία είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, πολύ πιο αμφιλεγόμενη από το θέμα των αμέσων πληρωμών. Έχω στο παρελθόν συγχαρεί την Κομισιόν για την πολύ καλή της πρόταση και βέβαια Παρ' όλα αυτά έχω καταθέσει και εγώ μια σειρά από τροπολογίες και οι συνάδελφοι έχουν υποβάλει σχεδόν 2.000 ε, τροπολογίες. Όλα αυτά είναι συμβολές οι οποίες είναι θετικές και τις περισσότερες από αυτές νομίζω ότι μπορώ να τις συμπεριλάβω στις συμβαστικές λύσεις στις οποίες θα καταλήξουμε. Εγώ κάνω αυτή τη στιγμή μια εξαντλητική εξέταση αυτών των τροπολογιών. Μπορώ να σας πω ότι περίπου το ίμιση από αυτές τις προτάσεις συνδέονται με το κεφάλαιο των μεμονωμένων μέτρων και πιστεύω ότι σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να ξεκινήσουμε την εργασία μας από αυτό το κεφάλαιο. Πρέπει να το πράξουμε αυτό, όπως κάναμε και στην έκθεση για τις άμεσες ε, πληρωμές, για να καθορίσουμε τη μέθοδο εργασίας μας και η μέθοδος εργασίας μας πρέπει να είναι παρόμοια με αυτήν που ακολουθήσαμε και στην άλλη έκθεση και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια θετική ε, λύση για τα θέματα αυτά. Συζητήσαμε για τέσσερις ώρες για το θέμα των άμεσων πληρωμών με πολύ θετικό πνεύμα από την πλευρά όλων των σκιωδών εισηγητών και μπορέσαμε με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουμε σε Συμβιβαστικέ τροπολογίε τι οποίε συζητήθηκαν στην Επιτροπή μα στη συνέχεια. Προτείνω και για αυτό τον κανονισμό να κάνουμε ακριβώ την ίδια διαδικασία και θα ήθελα να ακούσω προτάσει σε σχέση, για σε σχέση με τα θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε στην έναρξη της ε, ε, εξέτασή μα. Εγώ, όπω σα είπα προηγουμένω, προτείνω να ξεκινήσουμε με τα μεμονωμένα μέτρα που περιέχονται στι παραγράφου 15 έω 40 Δεν μπορούμε σε μία συνεδρία μόναχα βέβαια να εξαντλήσουμε όλο αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει το θέμα της μεταλαμπάδευσης ε, τεχνογνωσίας, παραγωγής συμβουλών, ε, επενδύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ε, επαναφορά της παραγωγικής ικανότητας μετά από φυσικές καταστροφές, τις βασικές υπηρεσίες στους Δήμους και τις κοινότητες, τις επενδύσεις στα δάση, υποστήριξη σε παραγωγούς, βιολογική γεωργία, ζώνες οι οποίες υφίστανται ειδική μεταχείριση. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει μια πληθώρα θεμάτων που όπως σας είπα ε, αντιστοιχούν σε περίπου 1030 τροπολογίες που είναι περίπου το ίμιση του συνολικού αριθμού τροπολογιών και επομένω, την Παρασκευή εμείς θα κάνουμε μια συνεδρίαση τεχνικού χαρακτήρα μεταξύ των συνεργατών των ε, συνεισηγητών και έτσι μπορούμε να έχουμε μια ημερήσια διάταξη για τη συνάντηση στις 26 Σεπτεμβρίου του εισηγητή με τους σκιώδους εισηγητέ. και εγώ θα σας πρότεινα να ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο αυτό ξεκινώντας από το άρθρο 15 και να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε για τα θέματα αυτά. <clears throat> Για τις τροπολογίες τώρα, σε γενικές γραμμές μπορώ να σας πω ότι το ΕΛΚ είναι αυτό που έχει καταθέσει τις περισσότερες τροπολογίες, 686 συγκεκριμένα. Και η δική μου ομάδα βέβαια. Άλλες 400 ε, πέραν αυτών που εγώ κατέθεσα ο ίδιος. Έχουμε φυσικά ένα τεράστιο πεδίο που πρέπει να εξετάσουμε, αλλά δεν μπορούμε φυσικά να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες μεμονωμένες, ακόμα είναι υπό επεξεργασία η ανάλυση τους. Εμένα θα με ικανοποιούσε να μπορούμε να έχουμε μια μέθοδο εργασίας που θα αποφασίσουμε σήμερα και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις και των άλλων πολιτικών ομάδων και φυσικά και πάλι θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και να εκφράσω την πλήρη διαθεσιμότητά μου για τι ανταλλαγέ απόψεων που είναι απαραίτητε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικέ συμβαστικέ ε, λύσει για ένα κανονισμό που είναι νευραλικός για το μέλλον των γεωργών και τη γεωργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ Λουί. Όπως συνηθίζεται, πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο στους σκιώδει ηγητέ και μετά τους σκιώδει ηγητέ θα ακολουθήσουν όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μιλήσουν. Elizabeth Kostinger και μετά Πόλσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή φυσικά θέλω να ευχαριστήσω για το έργο που έχει κάνει μέχρι τώρα και φυσικά και για την καλή συνεργασία που διατηρεί τις δυνατότητες μιας επικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας, όπως είπε και ο εισηγητής προηγουμένως, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των τροπολογιών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από τους διάφορους συναδέλφους και φυσικά είναι σημαντικές όλες αυτές οι τροπολογίες. Όταν κοιτάξει κανείς την τροπολογία έχει την εντύπωση ότι είναι ένας κατάλογος ονείων ή ένας κατάλογος ευχών και αιτήσεων προς τον Άι Βασίλη Είναι λοιπόν σημαντικό το να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και προτάσεις. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν διατυπωθεί αιτήσει για τα πάντα. Πρέπει επομένως για, σαν πρώτη προτεραιότητα να διαπιστώσουμε προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί η στοχοθεσία για την αγροτική ανάπτυξη, ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες, για ποια θέματα θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτές τις αιτήσει και ποιες είναι οι ομάδες στόχου τις οποίες πρέπει να υποστηρίξουμε. Και εδώ έχουμε ήδη κάνει επικοδομητικές συζητήσεις και νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητή είναι πολυθετική και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε θετικές συζητήσεις για όλα τα λεπτομεριακά θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινίσουμε μεταξύ μας. Εγώ νομίζω ότι οι έξι προτεραιότητες όπως έχουν παρουσιαστεί και οι οποίες αντικατοπτρίζουν σε κάποιο βαθμό την, τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί <clears throat> είναι ένας τρόπος εργασίας ο οποίος θα διατηρήσει και την ευελιξία στην εργασία μας και ο στόχος όλων μας πιστεύω ότι είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε τα προγράμματα επένδυσης και υποστήριξης, τα οποία είναι σημαντικά σημεία της πρότασης. Και επίσης ε, τονίζεται η ανάγκη να υπάρξει συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Όλες αυτές είναι λοιπόν βασικές προτεραιότητες και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για το πνεύμα συνεργασίας που έχει επιδείξει. Ευχαριστώ, Ελίζαμπεθ. Συνεχίζουμε. Αντιπρόεδρο Πόλσον. Με την Αντιπρόεδρο Πόλσον, Μαρία Πόλσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο Κάπουλο Σάντος. Έχω λοιπόν ε, μελετήσει όλες αυτές τις 2003 ε, τροπολογίες και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζουν όντως τις αντιδράσεις μας. Δεν είναι δυνατόν να μπερδευτούμε με όλες αυτές. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μέσα σε όλα αυτά. Συνεπώς πρέπει να προσπαθήσουμε στο κείμενό μας να βάλουμε προτάσεις και τροπολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις βασικές μας αρχές. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω τι πιστεύω εγώ ότι είναι η πιο σημαντική αρχή όσον αφορά την αναπτυξιακή μας πολιτική. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν θέλουμε να έχουμε μία γεωργία που να λειτουργεί και έναν δασικό τομέα που να λειτουργεί, τότε πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη μας και τα χωριά τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά στα δάση ή στα βουνά, είτε πρόκειται για ε, απομονωμένα στο βορρά ή στο νότο της Ευρώπης και που όμως έχουν έναν γεωργικό τομέα. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε να έχουμε έναν αγρότη που να είναι ευτυχισμένος από τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι στηρίζουμε και τις μικρές ε, επιχειρήσεις που προσφέρουν ε, αντίστοιχες υπηρεσίες για την γεωργία στα μικρά χωριά και τις πόλεις να λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική ζωή στον χώρο της υπαίθρου. Χρειάζεται, πρέπει να υπάρχει, γιατί μόνο αγρότες με οικογένειες μπορούν να επιζήσουν εκεί που δουλεύουν. Γι' αυτό το λόγο για μένα είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στην Ήπεθρο. Γνώση, ανάπτυξη γνώσης, μεταφορά γνώσης, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τους αγρότες στην Ήπεθρο. Τώρα, όσον αφορά τις λεπτομέρειες, θα έλεγα ας κοιτάξουμε τις δραστηριότητες μικρής κλίμακας. Η γεωργία από τη φύση της αποτελεί μία δραστηριότητα μικρής κλίμακας. Γιατί υπάρχουν ελάχιστες τεράστιες ε, κτηνοτροφικές, για παράδειγμα, εκμεταλλεύσεις γεωργικές. Ας δούμε και την δασοκομεία πολλοί κόσμος είναι υπέρ της δασοκομείας. Τάσετε υπέρ αυτής, αλλά σκεφτείτε λίγο τι γίνεται στα δάση στο βορρά της Ευρώπης. Δεν θέλουμε μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουμε ανώτατα επίπεδα. Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην δασοκομεία στην Ευρώπη βρίσκονται στον ε, Βορρά και δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιε τεράστιε επιχειρήσεις. Συνεπώ, ας μιλήσουμε για το ιδεώδες μέγεθο. Και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας για τον κόσμο της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Πόλσον. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σμιτ και θα χαιρετήσω και τους φίλους όμως που ήρθαν στην αίθουσα από τη Γερμανία, από τη Βόρεια Γερμανία, εκπροσώπους των διαφόρων ε, νόσων των περιφερειών. Καλώς ήρθατε όλοι. Και λέω ότι σήμερα το βράδυ στις 19.30 θα εγκαινιαστεί μια έκθεση που αφορά τα, προγράμματα αναπτύξεως ε, της, ε, της υπαίθρου της γερμανικής περιφέρειας. Συνεχίζουμε τον κύριο Σμιτ και μετά η Ελίζα Πεθιέγγελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Πολλοί από εμά νιώσαμε πολύ άνετα να συζητάμε μαζί του για τα διάφορα σημεία κλειδί της πρότασης. Ε, Όντω ήταν πάρα πολλές οι τροπολογίες που προτάθηκαν 2.000, από τις οποίες 120 ήταν από εμά Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για τις προτεραιότητές μας. Σας ελπίσουμε ότι και οι μεγάλες ομάδες να μπορέσουν να συντονιστούν τόσο καλά όσο συντονιζόμαστε κι εμείς. Τι να δεν μπορεί να τα έχει κανείς όλα. Έρχομαι όμως τώρα στην διαφορά φιλοσοφίας λιγάκι που υπάρχει για αυτό το θέμα. Όπως λέει και η κυρία Πόλσινγκ, πράγματι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι θέλουμε να πετύχουμε με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δυόμιση χρόνια ήμουνα στην Περιφερειακή Επιτροπή εδώ την κοινοβουλευτική, πέρασα εκεί δύσκολα χρόνια και ήταν ε, δύσκολο να το καθορίσουμε αυτό. Γιατί όταν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι σημαντικό να μην γίνει μια υπόθεση για την οποία όλοι μιλάνε και κανείς δεν κάνει τίποτα. Ήταν δύσκολο λοιπόν και στην Περιφερειακή Επιτροπή να προθίσουμε αυτό το θέμα. Πολλές ε, τροπολογίες θέλουν ε, αύξηση των ποσών, αλλά το θέμα είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου να ληφθεί υπόψη σαν κάτι που απαιτεί ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εκεί και των υποδομών. Σίγουρα θα συζητήσουμε για όλε τι τροπολογίε. Για μα το σημαντικό είναι η συγχρηματοδότηση. Εμεί θέλουμε μεγαλύτερο ποσοστό, 60% ενώ τώρα είναι 50% για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ή για την προστασία των ζώων. Υπάρχει η τροπολογία 9059 που αναφέρεται σε αυτά και στην συγχρηματοδότηση. Η δικιά μας τροπολογία 542. Ε, κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι πρέπει... Παρόλο που είμαστε ανοιχτοί στο οι αγρότες να μπορούν να μπουν σε ό,τι ε, εμπόρια, κερδοσκοπικά κτλ. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια δημόσιου χρήματο. Γιατί αυτό αποτελεί στρέβλωση. Την παραγωγή τροφίμων πρέπει να ενισχύουμε. Για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίε και εδώ είναι σημαντικό οι αγρότες να μπορούν να βοηθήσουν, να πάρουν μάλλον συμβουλές από αρμόδιους, είναι οι τροπολογίες μας 729, 734, 740 κλπ. Να λάβουμε υπόψη μας τις τοπικές ε, αγορές, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τον προπολογισμό τους πιο αποτελεσματικά οι αγρότες και αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο επίμαχο αυτό το θέμα. Θέλουμε στο άρθρο 20 να διαγράψουμε το πρόγραμμα που αναφέρεται εκεί. Είναι η τροπολογία μας 9.40 που πιστεύουμε ότι είναι σημαντική γιατί οι εγρότες αθαρρύνονται να βγουν από αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά τις συζητήσεις με τον εισηγητή για την ε, μεθοδολογία εργασία μας. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα αρκετά καλά. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στον προσανατολισμό μας ενδιαφέρουν. Ε, υπάρχουν οι συναντήσεις του προσωπικού, ή οι μόνο εγώ έχω υπογραμμίσω ότι τα άρθρα 15 με 40 πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη συζήτηση μας πριν προτείνουμε τον προπολογισμό. Εμείς θέλουμε ειδικά κείμενα να έχουν προετοιμαστεί και να έχουν μοιραστεί πριν από τις συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών για να μπορούμε πολύ συγκεκριμένα να συζητάμε πάνω σε αυτά. Ε, νομίζω ότι βλέπει κανείς από την συμπεριφορά της χειρονομής των άλλων ε, που θέλουμε να πάμε, αλλά μην είμαστε ντροπαλοί όμως, να έχουμε και κείμενα για να μπορούμε πολύ συγκεκριμένα πάνω σε αυτά να αποφασίσουμε. Από εκεί και πέρα προσδοκούμε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Τζαν Κάρλος Κότα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Δράτω σε ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον κύριο Καπούλα Σάντος για την έξοχη δουλειά που έκανε. Όχι μόνο στο θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου, αλλά και στις άμεσες πληρωμές. Η ανάπτυξη της υπαίθρου, κατά την άποψή μου, είναι η καρδιά, η παλόμενη της ΚΑΠ. Το λέω αυτό διότι τα μέτρα προβλέπονται εντό αυτής της πολιτικής θα πρέπει να ανταποκρίζονται στο πρόβλημα της περιφέρειας του Συνόδου της Υπέθρου. Αναφέρεται στις... Ε, συμφωνώ με τις απόψεις όσον αφορά τις περιοχές που έχουν ανάγκη υποστήριξη και άλλα θέματα. Η δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για δάνεια προς τους νέους γεωργούς σε κοινοτικό επίπεδο αυτό το μέτρο όχι μόνο μπορεί να υποστηρίξει αύξηση των νέων στον τομέα, αλλά πιο σημαντικά μπορεί να τους κάνει πιο υπεύθυνους και να τους δώσει κίνητρα στους νέους που θέλουν να πλησιάσουν την ύπεθρο και τον γυρικό κόσμο. Χωρίς να λάβουμε υπόψη αυτούς που διάλεξαν αυτή τη διαδρομή πρέπει να πολεμήσουν στεγαστικά δάνεια και τράπεζες υπό συνθήκες. Αν θέλουμε να γίνει ανανέωση των γενεών δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι θα πρέπει να ξανακαθορίσουμε ποιοι αποτελούν τους νέους γεωργούς. Πρέπει να τους δώσουμε σε αυτούς τους νέους όλα τα εργαλεία, τους ώστε επιτέλους να μπορέσουν να κινηθούν άνετα σε ένα τομέα τόσο σημαντικό ζωτική σημασία όπως είναι ο τομέας της γεωργίας. Ευχαριστώ Τζαν Κάρλο. Τελειώσαμε τους κοιόδους και τώρα συζητούμε με όλους συναδέλφους Ελίζαπεθ Γέγκελ και μετά ο Μισελ Νταντέν έχουν το λόγο. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πραγματικά εκ βάθους καρδίας τον εισηγητή του κύριο Κάπολο Σάντος για την εργασία που έχει ήδη φέρει σε πέρας και τις πολλές συναντήσεις που έχει κάνει και για τις προσπάθειες που έχει να καταβάλει και στο μέλλον. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει μια σωστή βάση εργασίας. Ίσως δεν κατάλαβα καλά αυτό το οποίο ακούσαμε από τους φιλελεύθερους. Αλλά δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η θέση των φιλελευθέρων. Ίσως θα μπορούσαν να διευκρινίσουν καλύτερα τη θέση τους. Α, η κυρία Πόλσεν. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τότε είμαι σε καλά χέρια με την κυρία Πόλσεν και εγώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή διαδικασία και είναι θεμητό το να υπάρχουν και τόσες πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και το ΕΛΚ έχει καταθέσει πιο πολλές τροπολογίες επειδή είναι η πιο πολυπληθής πολιτική ομάδα. Έχουμε ένα δύσκολο και κοπιώδες έργο μπροστά μας, αλλά είναι σημαντικό το έργο αυτό και αν μπορέσουμε εμείς να βρούμε τα κύρια σημεία τα οποία συνασπίζουν όλες τις πολιτικές ομάδες, τότε σίγουρα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Πιστεύω ότι είναι σωστό όλοι να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου είναι μια σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αγροτική ανάπτυξη έχει να αντιμετωπίσει και τις πιο μειονεκτικές και δύσκολες περιοχές και θέλω να τον τονίσω αυτό γιατί εγώ ακούω πολλές φορές φωνές αντίθετες στη χώρα μου. Τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να είναι για τους ε, αστικούς χώρους, αλλά θα πρέπει να είναι για την αγροτική ανάπτυξη. Οι χώροι των μεγάλων πόλεων, οι αστικοί συνασπισμοί, τα αστικά συγκροτήματα θα πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Και επίση δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη χωρί να λάβουμε υπόψη και τον, γυναικό, το ρόλο των γυναικών στι αγροτικέ περιοχέ. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό θα πρέπει να διατρέχει την έκθεσή μα, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλε τι ομάδε εργαζομένων στην γεωργία στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης και επομένως να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε οι περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ε, μειονεξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα προβλήματα να μπορέσουν και αυτές να επιβιώσουν. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή και όλους τους και εισηγητές και προβλέπω στη συνεργασία αυτών. Ευχαριστώ. Ο Μισελ Νταντέν και μετά Μπρίτα επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Κάτι που έχει σχέση και με τη δικιά μου έκθεση. Μιλάμε πολύ για το δεύτερο πυλώνα, για ό,τι έχει να κάνει με το πρασίνισμα ανάλογα βέβαια με τις ατομικές επιλογές του κάθε αγρότη. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες μελέτες που αρχίζουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας τελευταία και που δείχνει ότι τα 15 τελευταία χρόνια ο αγροτικός κόσμος αποτέλεσε αντικείμενο γενικά υποεπενδύσεων. Κάτι το οποίο εξηγεί σε ένα βαθμό τα προβλήματα παραγωγικότητας σε διάφορους κλάδους. Και αυτό τόσο στην έρευνα όσο και στον υπόλοιπο κλάδο. Έχουμε κλιματικές αλλαγές. Πώς θα διαχειριστούμε το θέμα αυτό, πώς θα διαχειριστούμε το θέμα του ύδατος και των αλλαγών που έχουμε στη βροχόπτωση. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε ελάχιστα συζητήσει στην Επιτροπή Γεωργίας. Αλλά αυτή η έλλειψη επενδύσεων που έχει λάβει η χώρα τελευταία γενικά στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει σύντομα. Ευχαριστώ, Μισελ. Μπρίτα Νέιμερ και μετά Μάρτιν Όσλιν. Μπρίτα. Ε, Ευχαριστώ και εγώ θέλω φυσικά καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο που έχει φέρει σε πέρας. Νομίζω ότι όλοι μας στην Επιτροπή μας πρέπει να συνεργαστούμε για μαζί του. Για μένα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο αυτό θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό του τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην Ήπεθρο και δεν μας ενδιαφέρει ένα αγροτικό ταμείο που έχει σαν στόχο να φύγουν από την Ήπεθρο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι όλα τα σχέδια τα οποία γίνονται για τον αγροτικό χώρο έχουν σαν στόχο να κάνουν τον αγροτικό χώρο ελκυστικό για τους εργαζόμενους και ζώντες εκεί. Δεν θέλουμε τα παιδιά των αγροτών να θέλουν να φύγουν και να πάνε στις πόλεις. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι επίση πρέπει να σκεφτούμε και μέσα στα πλαίσια της κρίσης του προπολογισμού που αντιμετωπίζουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της συγχρηματοδότησης. Εγώ αγωνίζομαι για το γεγονός να μπορέσει να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα ιδιωτική συγχρηματοδότηση στον αγροτικό τομέα. Γιατί υπάρχουν πολλέ περιφέρειε όπου είναι πολύ δύσκολο οι κυβερνήσει να εξασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση και θα πρέπει να βρούμε λύσει. Γιατί αλλιώ εν καιρό αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καθόλου επενδύσεις. Αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάσταση παράλογη <clears throat> την ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι και οι ασθενέστερε περιοχές θα εξελιχθούν εν καιρό για να φτάσουν το επίπεδο των πιο πλούσιων χωρών και περιοχών. Έχουμε πολλές θετικές εμπειρίες σε σχέση με τη συμμετοχή των αγροτών στην δική μας περιοχή. Αν συμμετέχουν σε μία εξέλιξη και σε, μια, σε κάποιο σχέδιο οι άνθρωποι εκεί, τότε θα το υποστηρίξουν και στη συνέχεια. Αλλιώς θεωρούν ότι γίνονται οι λήψεις αποφάσεων ερήμην τους και αυτό δεν τους οδηγεί να υποστηρίξουν. Εγώ νομίζω ότι αλλιώς αν συμμετέχουν έχουν και ένα πολύ θετικό αίσθημα σε σχέση με το ρόλο της Ευρώπης. Ο Μάρτιν Χάουσλινγκ και η κυρία Ρόντουστ μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα, βρισκόμαστε στο πραγματικό κάτω φράγμα, στο κάτω όριο αυτής της χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να συμπιέσουμε ακόμα προς τα κάτω τη χρηματοδότηση στον τομέα αυτό. Είπαμε και έχουμε τονίσει στο παρελθόν ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρονται κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα και θα πρέπει να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ώστε να είναι σε δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν στο δεύτερο πυλώνα. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς και αυτό είναι πρόβλημα για πολλά κράτη-μέλη που είναι η συγχρηματοδότηση όπως αναφέρθηκε. Αυτά τα οποία λέει η πρόταση Κομισιόν είναι σαφώς ε, χαμηλή χρηματοδότηση που θα οδηγήσει πολλά κράτη-μέλη σε προβλήματα για να συγχρηματοδοτήσουμε. Αυτό που αναφέρθηκε το θέμα της ιδιωτικής συγχρηματοδότησης για μένα είναι κάτι το οποίο αξίζει να το σκεφτούμε αλλά δεν μπορούμε να το δούμε σαν θεραπεία για το πρόβλημα αυτό γιατί πρέπει να σκεφτούμε από πού θα μπορούσε να έρθει το χρήμα του ιδιωτικού τομέα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως η λύση χωρί να εξετάσουμε την προέλευση αυτών των χρημάτων από το ιδιωτικό τομέα. Επίση έχουμε τα προβλήματα περιβάλλοντο στο δεύτερο τομέα, ε, τα οποία δεν υποστηρίζονται παρκώ ενώ συγχρόνω λέμε ότι θέλουμε το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα. Τα προγράμματα για το περιβάλλον στον δεύτερο πυλώνα είναι αυτά τα οποία προκρίνονται από τις περιφέρειες και μπορούν να συνδυάζονται με τα περιφερειακά προγράμματα. Δεν πρέπει να περιοριστούν τα προγράμματα αυτά. Κάτι άλλο το οποίο είναι σαφές είναι ότι στον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια να υποστηρίξουμε όχι μία ή δύο χώρες, αλλά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προκρίνουμε να υποστηρίξουμε τη βιολογική γεωργία. Κάτι άλλο το οποίο αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν είναι οι λεγόμενες ελάχιστες προδιαγραφές. Αυτό κινδυνεύει να κατεβάσει το επίπεδο προς τα κάτω σε χώρες οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες οι προδιαγραφές, ιδίως αν συνδυαστεί με τη χαμηλή χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε τα προγράμματα αυτά με διαφορετικό μάτι. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε σαφές στη συζήτηση ότι ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, ισότιμη μεταχείριση και όχι να καταλήγουμε πάντα σαν να είναι ο φτωχό συγγενή ε, του πρώτου πυλώνα, ο δεύτερο πυλώνα. Για μένα αυτό είναι το εργαλείο όπου μπορούμε, με το οποίο μπορούμε να κατευθύνουμε καλύτερα την ε, γεωργική πολιτική και να εκμεταλλευτούμε πολύ καλύτερα τις δυνατότητες που μας προσφέρει ο αγροτικός ε, χώρος για τη γεωργία και οι άλλες δραστηριότητε. Ευχαριστώ Μάρτιν. Ούλρικ Ρόλστρα και μετά ο Γκάμπλερ. Σας ευχαριστώ. Έχουν ελεχθεί πάρα πολλά που είναι σημαντικά στη συζήτηση και δεν θέλω να τα επαναλάβω όλα. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω τον Λοϊς Κάπολα Σάντος για την ευρύτατη και πλήρη εργασία του. Αυτά είναι θέματα που τα έχουμε συζητήσει διαμακρών στο παρελθόν του και έχουμε επομένως τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε σαφείς θέσεις. Εγώ πάντως θεωρώ ότι είναι γεγονός ότι πολλοί θεωρούν ότι ο δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να υποστηρίξει μόνο τη γεωργία και τίποτα παραπάνω. Για μένα ο δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να εξυπηρετήσει την τοπική οικονομία, την αγροτική οικονομία και ιδίως την συμμετοχή και την επιβίωση των ανθρώπων στον τομέα αυτό. Είναι ανόητο να θεωρούμε ότι αυτά είναι απλώς λεφτά που δίνουμε στους γεωργούς. Είναι μια τελείως λανθασμένη αντιμετώπιση. Για μένα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα ότι υπάρχει, ότι μπορούν να μεταφέρονται κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα. Αυτό είναι κάτι που έχει προταθεί όταν υπάρχει το λεγόμενο capping, δηλαδή το άνω όριο της χρηματοδότησης, τα χρήματα που περισσεύουν να πηγαίνουν στο δεύτερο πυλώνα. Όπως είπε και ο συνάδελφος Χόιστονγκ, η σκέψη για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδιωτικά ε, χρήματα για συγχρηματοδότηση και εγώ έχω διατυπώσει μια τροπολογία σχετικά, ξέρω ότι έχουμε πολλά ιδρύματα τα οποία μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο και με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την πίεση στα εθνικά κοινοβούλια και στα περιφερειακά κοινοβούλια. Φυσικά δεν θα πρέπει να ζητήσουμε ιδιωτική χρηματοδότηση χωρίς να ελέγχουμε από πού προέρχονται. Δεν θέλουμε να αναλάβουν τα ιδιωτικά συμφέροντα έλεγχο πάνω στη δραστηριότητα αυτά. Εμείς μας, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορούν οι περιφέρειες να είναι πιο ενεργέ στα θέματα αυτά και υπάρχει και μια έκθεση στο τρίτο πάτωμα από τη δική μου περιοχή, το Schleswig-Holstein, που δείχνει το πώς μπορεί μια περιφέρεια να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να έρθετε όλοι και να δείτε αυτή την έκθεση και θα διαπιστώσετε τι γίνεται με τα χρήματα του δευτέρου πυλώνα και πόσο σημαντικός είναι ο δεύτερος πυλώνας, επομένως και γιατί πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ουλρικέ. Χωρίς άλλο, δεχόμαστε την πρόσκλησή σου. Μαρία Γκάμπριελ και μετά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Καπουλάς ε, Σάντος και την ε, γραμματεία επίσης και να εκφράσω την ε, ελπίδα μου ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό τόπο στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε θέματα τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά για τη Βουλγαρία. Πρώτον, περιβαλλοντικά μέτρα. Πώς ορίζουμε ένα ελάχιστο ποσοστό. Πιστεύω ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να αποτελεί σύσταση και να μην είναι υποχρεωτικό. Διότι αν έχουμε ένα υποχρεωτικό τέτοιο μέτρο, τέτοιους δείκτες υποχρεωτικούς, τα κράτη-μέλη η κατάσταση διαφέρει. Οπότε τα μέτρα θα έπρεπε να είναι ελαστικά και να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με κλιματικούς και άλλους δείκτες. Επιτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες και να καθορίζονται τα ποσοστά και από την στρατηγική που υιοθετούν για τα περιβαλλοντικά μέτρα. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας είναι το εξής. Δασοκομεία. Εδώ υπάρχουν καταστάσεις όπου θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα εάν επεκτείναμε την εφαρμοσιμότητα των μέτρων αυτών, το παιδί εφαρμογή του δηλαδή. Στην Βουλγαρία είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε μια από τι λίγε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα δάση, όπου τα δάση κατά. σε ένα μεγάλο βαθμό ανήκουν στο κράτος. Πιστεύουμε ότι μέσα από το πρόγραμμα της υπαίθρου είναι δύσκολο να βρούμε χρηματοδότηση. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα πρέπει να απευθυνθούμε είτε σε ιδιώτες είτε στους δήμους ώστε να μπορούν να επωφεληθούν όλα τα δάση. Και να λάβουμε υπόψη μας και τις εταιρείες εκείνες τις κρατικές, οι οποίες όμως δεν εξαρτώνται άμεσα από τον κρατικό προπολογισμό. και να μειώσουμε βέβαια την ε, γραφειοκρατία. Και αν μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι που θα το υποστήριζα. Μαγκίνε τώρα. Και μετά ο αντιπρόεδρο ο Mm. Ευχαριστώ. Για... Ευχαριστώ τον εισηγητή. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μισελ Νταντάν για το ότι δεν υπάρχουν αρκετέ επενδύσει τελικά στην ε, Γεωργία. Πράγματι πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό καλό η κίνηση είναι αυτή η έκθεση. Τώρα συγχρόνω έχω και κάποιες ανησυχίε για τον περιορισμό των επενδυτικών ε, μέτρων όσον αφορά τις ε, ε, καλλιέργειες κάποιου μεγέθους και πάνω. Η χρηματοδότηση τώρα, ιδιαίτερα όταν συζητάμε για τον πυλήνα 1 το θέμα των άπεσων πληρωμών, εμείς έχουμε ζητήσει συγχρηματοδότηση η ομάδα μας. Βέβαια έρχομαι από μια χώρα που βρίσκεται σε πρόγραμμα λιτότητας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την άποψη για τη συγχρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να έχουν αποτελέσματα όλες οι χώρες, αλλά να ληφθούν υπόψη και τα προβλήματα κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Το άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Καταρχήν είναι μια καλή ιδέα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο μέτρο για τα κράτη-μέλη. Εδώ θέλω σχόλια από εσά. Δηλαδή πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο στην πράξη, πώς θα εφαρμοστεί. Η κύρια ιδέα πάντως που εγώ υποστηρίζω ένθερμα και από την αρχή την υποστήριξα, πρέπει να είναι Ας αναγνωρίσουμε λίγο περισσότερο την προσέγγιση, τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Για μερικά ε, κράτη-μέλη μπορεί να είναι κάτι που δεν χειρίζονται απευθείας μου τα κράτη-μέλη, αλλά να δίνουν αρμοδιότητες κι αλλού. Τώρα τα μέτρα πρασινίσματος από τον πρώτο πυλώνα που έχουμε συζητήσει και θα ξανασυζητήσουμε με τον εισηγητή έχουν επιπτώσεις και στον πυλώνα 2. Το γνωρίζετε, είμαι σίγουρη. Ας δείξουμε ευαισθητοποίηση εδώ και ας φροντίσουμε οι συζητήσεις να γίνονται παράλληλα και να μην ξεχνάμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο πυλώνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάριαν. Ο Αντιπρόεδρος ο και έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ίσως να μην πρέπει να μπούμε στη συζήτηση τη φιλοσοφική για τους πυλώνες αυτούς, αλλά το θέμα είναι ο δεύτερος πυλώνας είναι υπέρ της ανάπτυξης, είναι υπέρ του περιβάλλοντος ή πρόκειται για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στην πραγματικότητα, Γιατί όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να χρηματοδοτούνται από την κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις για να καταλάβουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν δαπανώνται απευθείας στη Γεωργία. Έμεσα ναι, αλλά όχι άμεσα. Πάνε στο περιβάλλον, Άρα ελάχιστα έχει να κάνει αυτό με τη γεωργία αυτή καθ' αυτή. Στο προήμιο πάντως λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν σε 25 με 30% το ποσοστό χρηματοδότησης για θέματα που έχουν να κάνουν με τις κλιματικές αλλαγές ή με την διαχείριση του εδάφους κλίμα, είπαμε, ε, άμεσες πληρωμές, οικολογική, γεωργία κλπ. κλπ. Οπότε, αυτό με οδηγεί στην εξή ερώτηση. Όλα αυτά είναι δεσμευτικά, είναι υποχρεωτικά ή όχι. Διότι κάπου αλλού στο κείμενο επαναλαμβάνεται το ίδιο, αλλά εκεί λέει θα έπρεπε να... Δηλαδή πράγματα τα οποία με κάνουν να πιστεύω ότι πρόκειται για υποχρεωτικά μέτρα. Και επιπλέον έχουμε και την οδηγία για το νερό, τα εφαρμοστικά μέτρα. καθώς επίσης και άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα. Οπότε η ερώτησή μου είναι Έτσι πρέπει να το διατυπώσουμε, σαν να είναι κάτι υποχρεωτικό ή βάσει της αρχής της επικουρικότητας να μην μένει ε, το πράγμα στα κράτη-μέλη. Και ποια είναι η ανάλυση η οικονομική αναπηλώνα Άλλοι δίνουν 40% στο δεύτερο πυλώνα και άλλοι δίνουν λιγότερα στο δεύτερο πυλώνα. Αν πάρουμε το 25% του 40% αυτού, αυτό κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ νομίζω ότι ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να πηγαίνει για την ανάπτυξη. Ένα άλλο θέμα, το οποίο βλέπω εγώ εδώ, είναι το θέμα εκείνο των ε, περιοχών που έχουν φτάσει στο 75% του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτή η αύξηση έχει επιτευχθεί από τόσα έχουν γίνει σε αστικό χώρο και όχι στην Ήπεθρο. Η Ήπεθρος αντίθετα δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα. Επιπλέον, όσον αφορά άλλα θέματα, θα τα δούμε βέβαια αργότερα, αλλά τέλος το μέγεθος του δεύτερου πυλώνα. Εδώ ακούμε ότι αν υπάρξουν περικοπές στον προπολογισμό, οι περικοπές αυτές θα γίνουν από το δεύτερο πυλώνα και την πολιτική συνοχής. Εγώ επιμένω ότι όταν μιλάμε για τη συνοχή, μιλάμε τελικά για τις πόλεις πιο πολύ και όχι για την ανάπτυξη της υπαίθρου ή ελάχιστα. Εγώ συμμετέχω και στην περιφερειακή πολιτική ως αναπληρωματικό μέλος. Μπορώ βέβαια να το συζητήσω εκεί, αλλά πιστεύω ότι αν θέλουμε να έχουμε αηφόρα ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, τότε τα χρήματα συνοχής πρέπει να πηγαίνουν και υπέρ της ανάπτυξης της υπαίθρου. Αν βέβαια θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Σεκεριέσκη. George Lyon και μετά θα δώσω στον Γενικό Διευθυντή Πλέβα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο. Απλώς σύντομα να πω κάτι και βασίζεται σε αυτό που μας είπε η Μαρία Μαγκίνες για την ε, εισαγωγή του κοινού στατικικού πλαισίου και για την χρήση των δικτών. Όταν η Επιτροπή Προπολογισμών συναντήθηκε με το Ελεκτικό Συνέδριο περίπου πριν από τετράμινο, αυτό συζητήθηκε εκτενώς και υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε, κυρίω από πλευρά Ελεκτικού Συνεδρίου. Δηλαδή, παρόλο που πίεζαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προ ένα σύστημα προσμέτρηση εκροή και όχι ζωή, αυτό που έχουμε τώρα Έχουμε και τα δύο συστήματα. Διότι όλες οι διαδικασίες ελέγχου επί της εισρωής που εστιάζονται επί της συμπληρώσεως των εντύπων και όλων των διαδικασιών ελέγχου θα εξακολουθούν υφίστανται ακριβώς όπως και προτέρω. Αλλά επιπλέον έχουμε τους δείκτες ε, εκροής. Δεν έχουμε ένα από τα δύο συστήματα, αλλά και τα δύο. Και αυτό είναι θεμελιώδες πρόβλημα που θα πρέπει να εξεταστεί. Είναι ξεκάθαρο και στην Επιτροπή Ρέτζη ισχύει αυτό γιατί είναι, αφορά την προσμέτρηση το, της χρήσης των πόρων και αφορά και την ρέτζη. Η Σκωτία συμμετείχε σε πολλά από αυτά τα ταμεία και κάποιε οργανώσει απομακρύνονται από τη χρήση του, διότι οι διαδικασίε ελέγχου είναι πάρα πολύ επαχθεί επί των διαφόρων φορέων. Και να προσθέτουμε τώρα και δείκτε εκροή ε, επιπλέον. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί τελικά μπορεί να κολλήσει το σύστημα και θα είναι πολύ δύσκολο να δαπανηθούν τα χρήματα λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα. Καλώ. ευχαριστώ Τζόρτζ. Σκέψη σημαντικότατη αυτή που εξέφρασες. Θα δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή Γιάννους Πλέμπα και μετά στον Λουίς για να ολοκληρώσει. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συγητή κύριο Κάπουλας Σάντους και τους σκιώδης εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για το τεράστιο έργο τους σε σχέση με το θέμα αυτό της αγροτικής ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο έχει προτείνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε αυτόν τον κανονισμό και η Κομισιόν το έχει καταγράψει. Πολλές από τις τροπολογίες και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου αφορούν τους στόχους και τις μελλοντικές προτεραιότητες αυτής της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και πολλές από αυτές τις τροπολογίες θα οδηγούσαν είτε σε μία υπερβολική διαστολή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ή θα την περιόριζαν ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να μην επιτύχει τους στόχους τους πραγματικούς αυτή η πολιτική. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εργαστούμε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Μια πολιτική που αντιμετωπίζει όλες τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η <clears throat> αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν συμμερίζεται την άποψη η οποία έχει εκφραστεί και σήμερα σε σχέση με την σημασία του δευτέρου πυλώνα στην αγροτική πολιτική. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να σχολιάσουμε τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία έχουν ε, τύχει της προσοχής των μελών της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά η μέθοδος εργασίας του εισηγητού είναι πολύ θετική και μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα, σε ένα ισορροπημένο τελικό αποτέλεσμα Το να ξεκινήσει λοιπόν η εξέταση του κανονισμού αυτού από τα άρθρα 15-40 μας φαίνεται ιδιαίτερα πραγματιστική. Θα περιοριστώ σήμερα στο να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ε, και τονίστηκαν ιδιαίτερα σε αυτή τη συζήτηση. Καταρχήν, για το ρόλο των κρατών μελών. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι χώρες μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συγχρηματοδοτούν κατά 25% τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των γεών και την, το μετριασμό των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής. Η Επιτροπή σας προτείνει μια συγχρηματοδότηση από, τα, από την Κομισιόν κατά 35, 40 ή και 50% παραπάνω. Αυτή η ηθική υποχρέωση δεν πρέπει να γίνει νομική υποχρέωση, ούτε πρέπει να καθοριστούν δεσμευτικά τα ποσοστά χρηματοδότησης. Η Κομισιόν θα δώσει περισσότερες εξηγήσει για τη θέση αν αυτό είναι απαραίτητο. Κάτι είναι σημαντικό σε αυτό το φάκελο είναι η αντιμετώπιση των περιοχών που έχουν φυσικά μειονεκτήματα. Για τις πληρωμές που αφορούν αυτές τις ζώνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει η μεταρρύθμιση να αναβληθεί μέχρι το 2015 και να αποτελέσει το αντικείμενο μιας χωριστής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ώστε και η θέση του Κοινοβουλίου να ληφθεί υπόψη, όπως και τα δεδομένα τα οποία θα υποβληθούν από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να προτείνω να υπογραμμίσω ότι η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες σε βάθος και που έχουν τύχει μίας ε, έχουν τύχει ελέγχου ομοτήμων όλες αυτές οι επιστημονικές μελέτες για κάθε μία από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση του Κοινοβουλίου οίκοθε εννοείται ότι θα ληφθεί υπόψη σε αυτήν την ε, έχει ληφθεί σε υπόψη σε αυτή την πρόταση. Γι' αυτό το να υπάρχει και χωρισμένη αντιμετώπιση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και η παρουσία μιας νέας νομοθετικής προτάσης που θα λάβει υπόψη αυτά τα, αυτές τις ανάγκες, χωρίς νέα στοιχεία θα καθυστερήσει χωρίς λόγο την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά. Τέλος, για τα προγράμματα leader τα οποία αναφέρθηκαν εδώ πέρα. Εγώ συμμερίζομαι την άποψη του Κοινοβουλίου σε σχέση με την οποία η προσέγγιση του leader είναι από τα κύρια μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να τονώσει τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο. μεταξύ των ταμείων λοιπόν που υποστηρίζουν τον αγροτικό χώρο, το Περιφερειακό Ταμείο είναι το μόνο του οποίου έχει καθοριστεί η ελάχιστη συμμετοχή για τα προγράμματα leader. Τα άλλα ταμεία δεν έχουν τέτοια κατώτατα όρια. Αυτό μας οδηγεί και σε μια συζήτηση για το αν τα κρατημέλη ή οι περιφέρειες θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα την κατεύθυνση του πρόγραμματος LIDER. Αυτό θα σήμαινε ότι το ελάχιστο επίπεδο θα παραμείνει στο 5% κάτι το οποίο σημαίνει ότι κανένα κράτος μέλος βέβαια δεν θα είναι δεσμευμένο να παραμείνει στο 5% θα μπορούσαν να δαπανίσουν <clears throat> περισσότερα ποσά. Είμαστε ως Κομισιόν έτοιμοι να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο επίπεδο της σε βάθος συζήτησης που θα ακολουθήσει μετά από τις συγκεκριμένες προτάσεις του εισηγητή. Καλώς, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Θα έλεγα, Λουίς, αν θες να εκφράσεις κάποιες τελικές σκέψεις, μάθεις υπόψη και τη σημαντική συζήτηση που διεξήχθη. Λουίς. Αγαπητέ Πρόεδρε, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα όλες τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων και που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτά που είχαμε πει σε διμερές επίπεδο τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες. Σίγουρα αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει μονάχα πολιτικό χαρακτήρα. Δίνουμε και την ψυχή μας και το συνέστημα στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τον αγροτικό χώρο και τη γεωργία. Δεν είναι όπως τα άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε μονάχα σαν πολιτικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάποια απόσταση και ψυχραιμία. Αυτά είναι θέματα που μας φέρνουν κοντά στις ρίζες μας και είναι συναισθηματικά θέματα, γι' αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας σημαντικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, μπορώ να υποστηρίξω τις περισσότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και καταγράφω αυτά τα οποία λέγονται. Παραδείγματος χάρη η ιδέα των ιδιωτικών επενδύσεων. Ξέρετε όμως ότι είναι σημαντικό οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα να υπόκειται πάντα σε ένα δημόσιο έλεγχο, μια αξιολόγηση από τις δημόσιες αρχές. Νομίζω ότι σε όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε σημεία ισορροπίας. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν. Βλέπω ότι υπάρχει ένα σημείο διαφοράς με την Κομισιόν που αφορά τον περιορισμό των περιοχών που θα την χάνουν υποστήριξη επειδή είναι μειονεκτικές. Αλλά εγώ περιμένω να υπάρξει συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές για να παρουσιάσω συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ Μέχρι στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ευρία ομοφωνία των σκιωδών εισηγητών που προσπάθησα να εξασφαλίσω ότι αντανακλάται και στην έκθεση. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθο και με την Κομισιόν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Η προστασία του περιβάλλοντος, οι αγροτοπεριβαλλοντικές προτάσεις, εκεί όταν προτείνω μια ελάχιστη χρηματοδότηση, αυτό έχει να κάνει με τη σχέση δεύτερου και πρώτου πυλώνα. Όπως ξέρετε, ο πρώτος πυλώνας είναι εκεί που εγώ προτείνω τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα να θεωρηθούν ως, ε, ως τη ούτα, υψοφάκτο δηλαδή, μέτρα πρασινίσματος. Και επομένως θα πρέπει να υπάρξει κατά την άποψή μου και μια αντίστοιχη αντιμετώπιση για τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα στον ε, δεύτερο πυλώνα που είναι και αυτά μέτρα για το greening. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια ελάχιστη ε, χρηματοδότηση για αυτά τα μέτρα για να είναι φανερό ότι εδώ δεν έχουμε μονάχα μια λεκτική δήλωση και απλώς λόγια, αλλά ότι είναι σημαντικά στοιχεία στην, στο πρασίρισμα της αγροτικής πολιτικής και εδώ πάλι θα αναζητήσω την καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση με την Κομισιόν. Συμφωνώ απόλυτα και με τον συνάδελφο Νταντά όταν μιλάει για το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην γεωργία μέσα στα θέματα έρευνας, ανάπτυξης και όλα αυτά. Όλα αυτά που έχουν χαθεί λοιπόν στον τομέα αυτό το, τα τελευταία χρόνια και βρισκόμαστε τώρα σε ένα νέο πλαίσιο, έχουμε νέες ανησυχίες για την τροφιμική ασφάλεια και την αυτάρκεια και για την ιδιαίτερη ε, πτυτικότητα των αγορών, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν τεράστιες διακυμάνσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην παρέμβασή μας και να έχουμε επομένω τα απαραίτητα μέσα και τους μηχανισμούς ε, ε, μεταφοράς κονδυλίων στον δεύτερο πυλώνα για την ενίσχυση αυτού του πυλώνα. Νομίζω ότι αυτά τα που έχουν προβλεφθεί μέχρι στιγμής είναι ανεπαρκή. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει και με, αναφέρεται και στην ε, έκθεση για τις άμεσες πληρωμές είναι ακριβώς αυτή η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των πυλώνων. Εγώ θα πρέπει να νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη μεταφορά κονδυλίων από τον πρώτο πυλώνα στην, ε, στο δεύτερο γιατί πολλά κράτη-μέλη έχουν μια αναντιστοιχία μέσων που δίδονται στον πρώτο πυλώνα και όχι στο δεύτερο θα πρέπει <clears throat> μέσα σε μια κατάσταση ύφεσης να αντιμετωπιστεί η μεγάλη δυσκολία που θα έχουν τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν επί κονδύλια στο δεύτερο πυλώνα, όπω είπε και ο συνάδελφο και υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ των δύο πυλών. Αν πάρω το παράδειγμα τη δική μου χώρα, είναι ε, μια κατανομή η οποία είναι σχεδόν ισόρροπη αλλά δεν ισχύει αυτό για όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτηση όλων των προτάσεων αυτών. Νομίζω ότι είναι καλό δεχτές όλες οι προτάσει. Υπάρχει ένα επικοδομητικό πνεύμα στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και ελπίζω ότι θα γίνει αποδεκτή η μέθοδο που εγώ έχω προτείνει να υπάρξει μια συνάντηση όπου θα καθοριστούν τα θέματα στα οποία θα υπάρξει ε, συζήτηση να δούμε πού είναι τα σημεία διαφορών και ποια είναι η διαδικασία να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις και θα σας ενημερώνουμε στο βαθμό που συνεχίζεται η συνεργασία των σχεδόν εισηγητών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε κάποιες θέσεις. Έχουμε χρόνο μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου που θα πρέπει να γίνει τελική ψηφοφορία και επειδή τώρα είμαστε σε μια, σε μια χρονική στιγμή που είναι ιδιαίτερα φορτωμένη η πολιτική διαδικασία, θα πρέπει να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες όλοι μας, αλλά όλα αυτά υπέρ της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Πολύ καλά. Ευχαριστώ, Λουί Κάπουλα Σάντο. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Γενικό Διευθυντή Πλέμπα. Η μέθοδο, ελπίζω, μα επιτρέψει να ξεφύγουμε από αυτό το μπλέξιμο των εκατοντάδων των τροπολογιών. Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 14 της σημερινής διάταξης, διότι το 13 Τζοβάνι Λαβία, ο συνάδελφος της Λαβία, είναι στην Επιτροπή Προπολογισμών και ζήτησε εάν θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε για μερικά λεπτά. Οπότε, αν ο Μάρτιν Όστενγκερ δεν έχει αντίρρηση, προχωράμε στο σημείο 14 ε, όσον αφορά τη μικροβιολογική πρόκληση, αυξανόμενος κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή. Θέλω να χαιρετήσω και την πολυπληθή αντιπροσωπεία των φίλων μα από την εκπροσώπων της Πούλια που είναι σήμερα. Τους χαιρετίζω όλους, Σέρβιο Μπράσβη, Αντώνιο Αντιάνη και όλους τους φίλους στην Επιτροπή Γεωργίας. Μάρτιν, σχέδιο δράση για την καταπολέμηση των αυξανωμένων κινδύνων όσον αφορά τι αντίσταση των μικροβίων, τη μικροβιακή αντοχή. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Σα υπενθυμίζω ότι με αυτή την έκθεση πρωτοβουλία η Επιτροπή μα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να τοποθετηθεί όσον αφορά το σχέδιο δράσης που θετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2011. Ο Μάρτιν Άστεγκερ είναι για την γνωμοδότηση και του δίνω αμέσως το λόγο. Μάρτιν, έχει το λόγο. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει προταχθεί το σημείο αυτό μεν, αλλά είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό και να λάβω το λόγο. Ξέρω ότι λαμβάνει χώρα μια τεράστια συζήτηση αυτή τη στιγμή για τα αντιβιωτικά στη Γεωργία και στη χώρα μου είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Και την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν στοιχεία για το πόσα αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται πραγματικά στη Γεωργία στην Γερμανία και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γενικά δεν έχουμε στοιχεία για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Αυτό είναι ένα από τα σημεία λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό πρότεινα τα κράτη-μέλη να έχουν μια μεγαλύτερη προσοχή για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συλλογή των στοιχείων για τα θέματα αυτά. Και βλέπω ότι έχουμε περίπου 1.700 τόνους ε, αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται στη Γεωργία 40 φορές παραπάνω από ό,τι χορηγεί ένα νοσοκομείο, ένα μέσο νοσοκομείο στην ε, Γερμανία. Αυτό σας δείχνει πραγματικά ποιο είναι, ποια είναι η έκταση του προβλήματος. 90% των ζώων έχουν ε, χορήγηση αντιβιωτικών. Η πρόταση της Κομισιόν πιστεύω ότι κινείται προς την κατεύθυνση που από τη σωστή κατεύθυνση, αυτό είναι σαφές, αλλά πιστεύω ότι δεν φτάνει αρκετά, δεν προχωράει αρκετά. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε για το θέμα αυτό, όχι μόνο με τα θέματα της έρευνας και για την ε, δημιουργία νέων αντιβιωτικών, αλλά θα πρέπει να δούμε καταρχήν να σκεφτούμε και να συζητήσουμε για το κατά πόσο το σύστημα εκτροφής ζώων είναι επαρκές και ε, σωστό και για το κατά πόσο θα πρέπει το σύστημα εκτροφής των ζώων το οποίο χρησιμοποιείται να οδηγεί μαθηματικά στην χορήγηση αντι, αντιβιωτικών σε όλα τα ζώα και αυτό πρέπει να είναι ένα σημαντικό θέμα στη συζήτηση που έχει να κάνει εναντίον της υπερβολικής χρήσης αντιβιωτικών. Και με τους σκιώδεις συζητητές νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας ότι τα αντιβιωτικά τα οποία βρίσκονται στους καταλόγους που ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας έχει θεωρήσει επικίνδυνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτά τα αντιβιωτικά να χρησιμοποιούνται έστω και περιστασιακά για την εξασφάλιση της υγείας των ζώων. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα λοιπόν το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε. Εγώ έχω συζητήσει λοιπόν εκ των προτέρων με τους σκιώδεις συγητές και έχουν τονίσει όλοι ότι αυτό είναι ένα κεφαλαιόδε σημείο. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ μας για τους σαφείς στόχους, όχι μόνο για τη χρήση αντιβιωτικών, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε μία εν καιρό μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών. Υπάρχουν χώρες όπως η Δανία όπου έχει μειωθεί κατά το ίμιση η χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Το θέμα δεν είναι μοναχά να κατανοήσουμε πώς αυτό είναι εφικτό, αλλά εμείς θεωρούμε ότι γενικά θα πρέπει να, να εξασφαλίσουμε μία μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών μέχρι το 2018 κατά 50%. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να θεσπίσουμε αυτό το στόχο και να τον κάνουμε δεσμευτικό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν με την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία όπως γίνεται. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην ε, κτηνοτροφία από τη χρήση αντιβιωτικών θα αντιμετωπιστούν. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, έχουμε συγκεκριμένους γεωργούς οι οποίοι κατηγορούνται για τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει όλος ο τομέας να αντιμετωπιστεί ως σύνολο. Θα είναι χρήσιμο επίσης τα μέτρα πρόληψης να παίξουν ένα σημαντικότερο ρόλο στην ε, συζήτηση. Όχι να θεωρούμε ότι τα αντιβιωτικά πρέπει να χορηγούνται συλλήδιν για προληπτικούς λόγους, και να υπάρχει μια συστηματική χρήση των αντιβιωτικών. Όταν έχουμε ένα ζώο λοιπόν το οποίο αρρωσταίνει σε μια αγέλη χιλιάδων ζώων δεν σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα ζώα θα πρέπει να ε, την χάνουν χορήγηση αντιβιωτικών. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο στοχευμένη αντιμετώπιση. Έχω μιλήσει και με τον εισηγητή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε και έχουμε ένα σωστό τρόπο αντιμετώπιση γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό ήδη υπάρχει συζήτηση σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά και ξέρουμε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία αν δεν αντιμετωπίσουμε με ενεργητικότητα το θέμα των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία και το να ακολουθήσουμε μονάχα την οδό τη Κομισιόν να έχουμε νέε μορφέ αντιβιωτικών, νέα φάρμακα, αυτό δεν υπάρχει. Πρέπει να έχουμε και μια πορεία προς τη μείωση τη χρήση των αντιβιωτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα γίνει η συζήτηση. Έχουμε την Αντιπρόεδρο Πόλσεν και μετά την Ελίζα Μπεθιέγγελ που θα μιλήσει. Η Μάριον Πόλσεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Συμφωνώ κατά 95% με τον εισηγητή. Ο τρόπος που περιγράφει την κατάσταση είναι ορθός. Τα στοιχεία είναι ορθά. Εγώ από τις αρχές ε, της δεκαετίας του 80 έχω αρχίσει να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Είναι τρομερό όμως που βλέπω ότι η κατάσταση σήμερα δεν έχει αλλάξει καθόλου από ότι τότε όταν άρχισα να ασχολούμαι. Αντίθετα, επιδεινώνεται θα έλεγα κάθε χρόνο. Την δεκαετία του 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε την απόφαση τα αντιβιωτικά να μην χρησιμοποιούνται για, να... για την πάχυνση, για παράδειγμα, αλλά προφυλακτικά. Τα αντιβιωτικά όμως τελικά σήμερα χρησιμοποιούνται περίπου με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και είναι κάτι που μας αφορά όλους. 70% περίπου όλων των ασθενειών που αντιμετωπίζονται με αντιβιωτικά ε, απαντώνται όχι μόνο στο ανθρώπινο είδος αλλά και σε πολλά άλλα θαλαστικά. Και 98% περίπου για να μην πω 100% των ε, ασθενειών που οφείλονται σε βακτηρίδιο και πλήττουν ε, τους χείρους ε, πλήττουν και τους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν θα έπρεπε, πιστεύω, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται σήμερα τα αντιβιωτικά. Δηλαδή, σε ποια συστήματα κτηνοτροφίας χρησιμοποιούνται, σε ποια είδη ζώων πρόκειται για τα βοηδή, τους χείρους και γεωγραφικά να έχουμε επίσης μια χαρτογράφηση της κατάστασης. Και εκείνο που δεν συμφωνώ με τον κύριο Χόισλινγκ στο ότι δεν είναι θέμα μόνο ποσότητας, είναι θέμα τι είδους αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε μια πρόταση που λέει ότι τα τέσσερα πιο αποτελεσματικά αντιβιωτικά που έχουμε σήμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική. Αυτά τα τέσσερα είδη αντιβιωτικών που είναι τα πιο αποτελεσματικά θα πρέπει να περιορίζονται μόνο για ανθρώπινη χρήση. Συνεπώς, δεν μπορεί να φτάνει η συνταγογράφηση από έναν κτηνίατρο, θα πρέπει να χρειάζονται δύο κτηνίατροι για να ζητήσουν ένα τέτοιο φάρμακο. Είμαστε δηλαδή σήμερα σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα. Έχω συνεργαστεί με τον εισηγητή και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του. Και θα ήθελα μια πιο συγκεκριμένη πρόταση για τη χρήση των αντιβιωτικών. Η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία έχει έχουν ένα αξιοπρεπές σύστημα ελέγχου των αντιβιωτικών. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να βασιστούμε στα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Είναι συστήματα τα οποία δεν είναι τόσο γραφειοκρατικά για τους αγρότες και δεν πρέπει να είναι, αρκετή δουλειά έχουν με τα γραφειοκρατικά. Οι κτηνίατροι πρέπει να κρατούν στοιχεία για τις διαγνώσεις που κάνουν στοιχεία τα οποία πρέπει να συλλέγονται μαζί και έτσι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης. Ενώ σήμερα δεν έχουμε ιδέα για το τι συμβαίνει περίπου. Ευχαριστώ κυρία Πόλσον. Ελίζα Πεθ Γέγκελ και μετά Μπρίτα Ρέιμας. Η Ελίζα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την προλαλήσαντα, την προλαλήσασα την κυρία Πάουσεν. Όπως είπε η κυρία Πάουσεν, είναι σωστά αυτά που είπε η κυρία Πόλσεν και αυτά που Είπε ο κύριο Χόισλινγκ, τα υποστήριζω αυτά που γράφει όμω στην εκθεσή του, δεν μπορώ όλα να τα υποστηρίξω. Η κυρία Ρόσπαχ από την Επιτροπή Περιβάλλοντο, που είναι η αρμόδια επί τη Επιτροπή, έχει κάνει μια πολύ καλή έκθεση. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να υποστηρίξουμε αυτά που λέει η κυρία Ρόσπαχ, η οποία έχει ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα αυτό. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και το τόνισε ο κύριο Χόισλινγκ για τη γεωργία. Η γεωργοί πρέπει να τεκμηριώνουν τη χρήση των ε, αντιβιωτικών, αλλά αυτό δεν ξεπενάει απλώς τη συνταγογράφηση αυτών των ε, φαρμάκων. Αυτά τα οποία αναφέρατε για τη χρήση ε, αντιβιωτικών στην γεωργία ε, είναι εντυπωσιακά. Αλλά εδώ έχουμε τα ζώα τα οποία χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα ζώα, αλλά είναι και τα ζώα τα κατοικίδια τα οποία επίσης λαμβάνουν αυτά τα αντιβιωτικά. Για μένα το σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μια σαφή τεκμηρίωση το πού πηγαίνουν τα φάρμακα αυτά, τα αντιβιωτικά. Έχουμε ζητήσει στη Γερμανία εδώ και από πολύ καιρό να υπάρχει σωστή παρακολούθηση των αντιβιωτικών και αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η κυρία Ρέσβαχ. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει μια σωστή έκθεση και πρέπει να την υποστηρίξουμε και γι' αυτό η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας δεν πρέπει να ξεπεράσει τα εσκαμένα και να αλλάξει το χαρακτήρα αυτής της έκθεσης της ε, κυρίας ε, Ρόσπαχ. Γι' αυτό θέλω να πω στον κύριο Χόισλινγκ ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω το, τη γνωμοδότησή του με όλα αυτά. Η, η Μπρίταρ και η Μαρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ λέει η κυρία Ρέμες. Και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Κάτι το οποίο με τρομάζει είναι ότι ενώ έχουμε τον ίδιο στόχο φαίνεται κάπου να υπάρχει μια προσπάθεια προεκλογικής εκμετάλλευσης. Ξέρω ότι οι πράσινοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κτηνοτροφία ως ένα από τα προεκλογικά τους θέματα και εμείς θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το που υπάρχουν οι διαφορές. Ο κύριος Χόισλιν κάνει μια σύγκριση μεταξύ της χρήσης αντιβιωτικών στα νοσοκομεία και για, την, ε, για τα ζώα, αλλά δεν κάνει διάκριση μεταξύ των ζώων τα οποία εκτρέφονται και των ζώων που είναι κατοικίδια. Δεν λέει κανείς ότι ακόμα και στα νοσοκομεία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αντιβιωτικών τα οποία δίδονται χωρίς πραγματικό έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε όταν συζητάμε για αυτό το θέμα το οποίο είναι ένα θέμα του μέλλοντος με να έχουμε σωστά στοιχεία. Πρωτού αρχίσουμε να καταδικάσουμε επί τη βάση στοιχείων τα οποία δεν είναι τεκμηριωμένα, κάτι το οποίο δεν συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι και τα ζώα έχουν το δικαίωμα για την θεραπεία με αντιβιωτικά όταν τα χρειάζονται. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μια αντιμετώπιση συλλήβδην εναντίον αυτών των πραγμάτων. Επίσης έχουμε διαφορετικές ενεργές ουσίες. Οι διαφορετικές ουσίες αυτές έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τη χρήση αντιβιωτικών στα ζώα με τη χρήση αντιβιωτικών στα, στους ανθρώπους. Και αναφέρεται επίσης ότι έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκτινοτροφία. Γιατί ε, βλέπω ότι δεν έχει να κάνει με τον τρόπο εντατική ή κτηνοτροφίας όπως δείχνουν οι μελέτες. Πολλές φορές ο μεγάλος αριθμός ζώων μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη προστασία τους. Γι' αυτό όπως έχει η έκθεση και εγώ δεν μπορώ να την υποστηρίξω Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο για τα θέματα αυτά και πώς μπορούμε να κινηθούμε για να υποστηρίξουμε καλύτερα την έκθεση της κυρίας Ρόσμπαχ, η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική έκθεση. Νομίζω λοιπόν όμως ότι η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να κάνει μικρές βελτιώσεις στην έκθεση Ρόσμπαχ, αλλά γενικά να την υποστηρίξει και όχι να στραφεί εναντίον της. Ευχαριστώ Μπρίτα. Μαρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Η κυρία Πόλσον, η κυρία Γέγκλερ, η κυρία Έμες, όλοι μίλησαν για αυτά που θα μιλήσω κι εγώ, συμφωνώ μαζί τους. Συμμετείχα και στη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και υποστηρίζω ότι η έκθεση Ρόσπακ είναι καλή. Με κάποιες τροπολογίες θα ήμουν ευτυχής. Ο κίνδυνος που ελοχεύει εδώ είναι να βάλουμε σαν στόχο ένα νούμερο χωρίς να βάζουμε καμία απόχρωση για τις συνέπειες κάτι τέτοιο. Το θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης που προστίθεται είναι κάτι που δεν θέλω. Συμφωνούμε με το στόχο όλοι. Και ίσως διαφέρουμε ως προς το πώς θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Και υπάρχει, πιστεύω, μια υπερβολική αντίδραση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε την κατάληξη που θέλουμε. Ο συνάδελφος κ. Χαλφίν είπε ότι ότι τελικά το πρόβλημα είναι οι μήκητες στα νοσοκομεία που προκαλούν ε, ε, μολύνσεις. Και στα κράτη-μέλη το ξέρει αυτό ο ιατρικός κόσμος, οπότε ο καλύτερος τρόπος να το αποφύγουμε είναι η σωστή υγιεινή. Έτσι προστατεύουμε τον άνθρωπο. Σημερίζω λοιπόν λέγοντας ας δούμε τι έχει κάνει και η Επιτροπή ΕΝΒΗ, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και έτσι να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που συνδέεται με την πραγματικότητα περισσότερο. Περισσότερο με αυτό από άλλε πτυχέ που θα μπορούσαν να πειράσουν τη συζήτησή μα. Ευχαριστώ του συζητητέ, ευχαριστώ τον Μάρτιν. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να είναι από τη Γενική Διεύθυνση Υγεία, DG Sanko, κάποιο εκπρόσωπο. Ποιο θα πάρει το λόγο. DG Mr. Van Dijk. Ο κύριος Βαντίκ ή ο κύριος Δεσμέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, όπως γνωρίζετε και από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μικροβιακή αντίσταση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίστηκε σαφώς στην έκθεση που θετήθηκε το Νοέμβριο του 2011 και όπως προαναφέρθηκε από αρκετούς προλαλήσαντες, ήρθε η ώρα για συγκεκριμένες πράξεις και στην έκθεση αναφέρεται στο σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα δείτε το σχέδιο δράση αναφέρεται σε συγκεκριμένε δράσει για την αντιμετώπιση τη απειλή τη μικροβιακή αντίσταση. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω, κάτι που αναφέρθηκε, είναι η σημασία να ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση. Όταν μιλάμε για τη μικροβιακή αντίσταση, δεν μπορούμε να δακτυλοδεικτούμε έναν τομέα ή μία πλευρά της αλυσίδας, αλλά πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται από πλευρά ανθρώπινης υγείας και υγείας των ζώων. Σημαντικότατο λοιπόν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όλοι οι φορείς και πλευρά της υγείας των ανθρώπων και της υγείας των ζώων να συμβάλλουν όλοι για την καταπολέμηση της αντίστασης των μικροβίων. Τώρα έρχομαι σε πιο συγκεκριμένα σχόλια. Πρώτα απ' όλα κάτι που συνδέεται με τη σχέση των πολύ της κρισίμου σημασίας αντιβιωτικών και στην αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα αυτό είναι κάτι θα ληφθεί υπόψη και θα εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς το θέμα των κρισίμου σημασίας αντιβιωτικών και αν θα πρέπει ε, να εξαιρούνται στην κτηνοτροφία ή να μην εξαιρούνται. Να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων στο Λονδίνο να εξετάσει τον αντίκτυπο που έχει τη δημόσια υγεία η, η χρήση αυτών των κρισίμων αντιβιωτικών στην ε, κτηνοτροφία. Θα δοθεί λοιπόν αυτή η εντολή στην ΕΜΕΑ, ούτως ώστε να εξετάσει εκ του στο θέμα. Το άλλο, σωστή συνετή χρήση. Και αυτό είναι ένα θέμα που επί μακρόν συζητείται, η συνετή προσεκτική χρήση και σχετικά με αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για νομικές διατάξεις για την υποστήριξη της ενίας αυτής. Πέραν αυτού, εν αναμονή μελλοντικών ενδεχομένων νομικών αλλαγών, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη επί καλών παραδειγμάτων για να αναπτύξουμε ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς για τη συνετή χρήση. Έτσι θα βοηθηθούν τα κράτη-μέλη που ίσως είναι λιγότερο προχωρημένα, τόσο ώστε να ωφεληθούν από τη γνώση των πιο προχωρημένων κρατών και να βοηθηθούν από προσανατολισμού για τη συνετή χρήση των ουσιών αυτών στην κτηνοτροφία. Έλεγχο, ενημέρωση, υποβολή εκθέσεων. Βασικά θέματα τα ανέφεραν και τα μέλη. Βασικό στοιχείο όταν μιλάμε για την ε, αντίσταση των μικροβίων. Δεν μιλάμε για τη χρήση των αντιβιωτικών, από πλευρά κτηνιατρική αλλά και πλευρά ανθρώπινη υγεία ξεκινήσαν προσπάθειες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που εξετάζει την χρήση, την χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. 20 κάτι μέλη συμμετέχουν. Αναμένεται έκθεση το τέλος 2012. Θα αναφέρεται συλλογή στοιχείων σχετικά με τη χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Το έγγραφο αναμένεται τέλος 2012 όπως προανέφερα. Κάτι άλλο σημαντικό. Όχι μόνο χρήση αντιβιωτικών, αλλά έλεγχος της αντιστάσεως των μικροβίων. Αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε το όφελος των δράσεων που εφαρμόζουμε. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είδατε ότι δεν αναφέραμε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο όσον αφορά τη μείωση του προβλήματος. Θέλουμε μέσω εναρμονισμένου ελέγχου να δούμε κατά πόσο τα μέτρα είναι αποτελεσματικά μετά από πέντε χρόνια. Και γι' αυτό ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλεία Τροφίμων να εξετάσει και να μας συμβουλεύσει για την καλύτερη προσέγγιση, τα καλύτερα κριτήρια που θα μπορούσαν να συμμεριληφθούν στην, στην εναρμονισμένη υποπτία, εν κατακλείδη. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υψή τη σημασία και προτεραιότητα στο θέμα, θέλουμε να κινηθούμε και στο νομικό τομέα, μέσω νομοθεσία, μέσω κατευθυντηρίων γραμμών, αλλά υποστηρίζουμε πλήρω την προσοχή που δίδεται στην αντίσταση των μικροβίων από πλευρά Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαντίκ, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ξαναδίνω το λόγο στον Μάρτιν για τα συμπεράσματα. Έχει το λόγο, Μάρτιν. Ähm, Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω για τι παρεμβάσει σα και τη συμβολή σα στη συζήτηση. Προσπαθήσουμε φυσικά να επεξεργαστούμε όλες αυτές τις προτάσεις, αυτό είναι σαφές για την κυρία Ρέματς και την κυρία Γέγκλα. Ε, τώρα, το θέμα που αναφέρατε για τον προεκλογικό αγώνα στη Γερμανία το βρίσκω κάπως ε, παράλογο. Εγώ αναφέρθηκα σε στοιχεία του Υπουργείου Υγείας στο, από την ε, Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Έχουμε μια αύξηση από το 2005 750 τόνων περίπου. Δεν χρειάζεται να παίζουμε παιχνίδια. Δεν πρόκειται για τις γάτες και τους σκύλους τα κατοικίδια ζώα. Πρόκειται για τα ζώα τα οποία εκτρέφονται στι ε, κτηνοτροφικέ εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ακόμα και αν υπάρχει το θέμα αυτό στη Γερμανία αυτή τη στιγμή που είναι επίμαχο, σίγουρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τη κτηνοτροφία. Υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να είμαστε και επικριτικοί εν ανάγκη. Πρέπει να σκεφτούμε και την ε, επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία που αυτή τη στιγμή είναι αδιαμφισβήτητη και μας δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες ότι κάποια στιγμή τα αντιβιωτικά πάβουν να λειτουργούν λόγω ακριβώς αυτής της υπερφόρτωσης αντιβιωτικών στα ζώα εκτροφής. Δεν πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Σας έκανα σαφής, σαφές αυτά τα, σε αυτά που είπα ότι μιλάω για τάξεις μεγέθους για, στη χρήση των ε, αντιβιωτικών και στην ε, χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα εκτροφής και όλα αυτά τα έχουν δείξει μελέτες στη Γερμανία και στα διάφορα κρατήδια της Γερμανίας. Όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, δεν πρέπει να τα αποφύγουμε και πρέπει να αφήσουμε τα, να τονίσουμε τη σημασία αυτών των θεμάτων. Η πρόταση της κυρίας Ρόσπαχ είναι σωστή από την Επιτροπή Γεωργίας, λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρει και πρέπει να είμαστε όμως λίγο πιο σαφείς στα θέματα αυτά. Το να υπάρχει μια τεκμηρίωση για τα αντιβιωτικά και τη χρήση των αντιβιωτικών, αυτό από μόνο του δεν οδηγεί στην μείωση της χρήσης αντιβιωτικών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρώπη για να μειωθεί η χρήση των αντιβιωτικών. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι κατευθύνσεις μπορούμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να υποβαθμίσουμε τη σημασία αυτού του θέματος, πρέπει να επιληφθούμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Μάρτιν. Σου εύχομαι να συνεργαστείς άριστα με τους κοιόδης ηγητές, ούτως ώστε να κατορθώσεις να λάβεις υπόψη ποια θα είναι η πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση. Τα στοιχεία της Γερμανίας είναι σημαντικότατα προφανώς αλλά θα πρέπει να δώσουμε μια έκθεση πρωτοβουλία στην γνώμη μα όσον αφορά την κατάσταση στην Ευρώπη και είμαι σίγουρο με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να το πετύχουμε. Υπενθυμίζω στου συναδέλφου την προθεσμένη υποβολή τροπολογιών όσον αφορά την έκθεση του Μάρτιν Άστεγκερ που είναι αύριο 19 Σεπτεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Είναι σημαντικό για όποιον θέλει να υποβάλει τροπολογίε. Αύριο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία. Έφτασε ο κύριο Λαβία Πάμε στο σημείο 13, διότι ήταν στην Επιτροπή Προπολογισμών. Είμαστε στο τέταρτο θέμα που αφορά την μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική, χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση τη ΠΑΚ, τη κοινή γεωργική πολιτική. Το λόγο έχει εσύ, Τζοβάνι, και μετά ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή Μέγκελ τη DG Agri ε, για την παρουσία του, που μετά θα πάρει το λόγο να μα μιλήσει. Ο Τζοβάνι, καταρχά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο οριζόντιος κανονισμός προφανώς είναι ένας από τους κανονισμούς εκείνους που συνδέεται με όλους τους άλλους, οπότε έχουμε μεγάλη εξάρτηση και από τις άλλες εκθέσεις οι οποίες συζητούνται από αυτήν την Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο αυτό. Επιτρέψτε μου να προβώ σε συντομότατη εισαγωγή για να δώσω μετά περιθώριο στους συναδέλφους να μιλήσουν και να ακούσω προσεκτικά τα σχόλιά τους. Είναι σαφές ότι όσον αφορά τους άλλους εισηγητές σχέση με τους άλλους πρέπει να θεωρώ στον εαυτό μου τυχερό διότι πήρε, έλαβα μόλις 648 τροπολογίες οπότε η δουλειά μου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι πιο εύκολη σε σχέση με τα όρια που έπρεπε να, στα οποία έπρεπε να ρηχηθούν οι συνάδελφοι, στα όρια των τροπολογιών. Ε, οι τροπολογίες όμως που για τις άλλες εκθέσεις έχουν και ε, επιρροές στη δική μου. Θα έπρεπε να τα εξετάσουμε όλα αυτά μαζί για να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στην όλη διαδικασία της συναπόφασης που ε, μας κάνει να προσπαθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μετά σε συζητήσεις στο Συμβούλιο επιλογές που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι και οι πιο χρήσιμες για τη Γεωργία και για τους Ευρωπαίους Γεωργούς και για την Ήπεθρο βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε σε ένα προβληματισμό όσον αφορά τους βασικούς άξονες, τα βασικά στοιχεία που είναι επίμαχα στην έκθεση αυτή και σε εκθέσεις αυτές και να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποια σημεία επί των οποίων επικεντρώθηκε η προσοχή των συναδέλφων και σε κάποιες περιπτώσεις βλέπω να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση σε κάποια σε, άλλα σημεία υπάρχουν διαφορές. Και θα πρέπει να συζητήσουμε επ' αυτών για να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι μια πρόταση ε, συμβιβαστική. Για να δώσω κάποια παραδείγματα, θα εστιάσω την προσοχή μου επί κάποιων θεμάτων. Εν πρώτης, το άρθρο 12, το σύστημα για τη διαβούλευση με τις επιχειρήσεις, όπου εκεί Λάβαμε 59 τροπολογίες και υπάρχουν ακραίες θέσει που συμπεριλαμβάνονται που θέλουν να εξελίψουν αυτό το σύστημα κάποιες αλλά οι τροπολογίες των συναδέλφων εστάθηκαν περισσότερο επί των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα πρέπει να εφαρμόζει αυτή η υπηρεσία και ποιοι θα πρέπει να είναι δικαιούχοι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία θέσεων και θα πρέπει στη συζήτηση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στο οποίο συμφωνήσαμε με τους κοιόδης, θα πρέπει να συζητήσουμε λέγω και να εστιαστούμε επί κάποιων σημείων αυτών των σημείων και να βρούμε έναν ελάχιστο κοινό συντελεστή. Δεύτερο θέμα είναι της ε, ρεσιμότητας. υπάρχουν και διάφορες ερωτήσεις που απορρέουν από τις τροπολογίες. Ποιος θα πρέπει να εξαιρείται από το καθεστώς. Ε, κάποιος ε, λέει ότι το καθεστώς θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους εκείνους που χρησιμοποιούν τις ενισχύσεις τις άμεσες της κοινή αγροτικής πολιτικής. Άρα ότι δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν οι μικροί καλλιεργητές διότι αλλιώς ε, υπάρχει στρέβλος ανταγωνισμού και δεν υπάρχει συνοχή στην πρόταση. Κάποιοι άλλοι λένε αντιθέτως ότι πέρα από τη διάσταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κάποιων τομέων της γεωργίας κάποιοι που ενδιαφέρονται και κάποιοι που δεν ενδιαφέρονται τόσο. Ε, και αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε. Άλλο ευαίσθητο θέμα είναι το σεβασμού της οδηγίας για τα ύδατα, διότι είναι προφανές ότι θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να απορρεύσουν από ενδελεχή συζήτηση σε κάποιο άλλο βήμα. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μέχρι το 2014 κάποια διέξοδο βλέποντας τη μεγάλη ποικιλία των θέσεων όσον αφορά την ευρωπαϊκή θέση και να υπάρξει και συνεννόηση. Η εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα και η λήψη υπόψη αυτής στην ερεσιμότητα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το θέμα των διπλών πληρωμών. Προτείναμε να διευρυνθεί δυνατότητα να εισπράκτει κανείς την πληρωμή από το πρασίνισμα και για εκείνους που εφαρμόζουν αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Πέραν από εκείνο που κάλυπτε η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εφάρμοζαν την ε, βιολογική παραγωγή. Αλλά από κανένα συνάδελφο όμως δεν έφτασε κάποια πρόταση όσον αφορά τη συμπερίληψη εκείνων που λειτουργούν στις περιοχές Natura 2000. Ε, περίμενα κάτι από αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έφτασε κάτι. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Το θέμα του διαχωρισμού των κυρώσεων όσον αφορά, ε, μάλλον του διαχωρισμού βασικών πληρωμών από τι πληρωμέ για το πρασίνισμα. Δύσκολο να δούμε ποιο συμμορφώνεται και ποιο συμμορφώνεται. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Μετά έχουμε το θέμα τη ευθυγράμμιση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πακέτο τροπολογιών που συνάδουν εν με την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τοποθετήθηκε επί τη ευκαιρία των συζητήσεων για την ευθυγράμμιση του πρώτερης ρυθμίσεως πριν από τη συνθήκη της Αβώνας. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν και διαφορετικές θέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συζητηθούν. Μετά έχουμε άλλο θέμα της απλούστευσης. Πρέπει να πω ότι σε όλη την Ευρώπη και στι διάφορε συναντήσει που είχαμε στην Ευρώπη, κάποιε προτάσει που με ικανοποίησε περισσότερο, μάσε περισσότερο, είναι αυτή που ήταν εντό τη έκθεση για την απλούστευση. Δυνατότητα για πολιτεί αιτήματα, αιτήσει για να μειωθεί η γραφειοκρατία για του γεωργού. Και επ' αυτού υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει. Και αν υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, θα πρέπει να συζητηθούν για να βρούμε λύση. Μετά είναι θέματα που αφορούν τι λεπτομέρειε. του τύπου πώς οι λεπτομέρειες των ελέγχων. Και οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν τόσο και από μικρές περιοχές. Οι περιοχές του πρασινίσματος Φερρυπίν. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας λεπτομερή χαρτογράφηση των περιοχών ε, και εδώ υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και υπάρχει χρόνος και περιθώριο και επ' αυτών να επιτευχθεί η συμφωνία. Θεωρώ σημαντικό να υπογραμμίσω και ίσως είναι το σημαντικότερο αυτό, τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, που είχα υπόψη μου. Προγραμματίσαμε την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο βοηθών για να ξεκινήσουμε μια εξέταση των απόψεων, να δούμε που αποκλίνουν. Μια πρώτη συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές προβλέπεται για τις 3 Οκτωβρίου και μετά μια έκθεση με βάση τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν υπάρξουν, που θα έπρεπε να υπάρξουν, και να δούμε αν υπάρχει ανάγκη συνέχισης των συναντήσεων, εάν σύντομα μπορούμε να βρούμε μια πλήρη γενική συνεννόηση μεταξύ πολιτικών ομάδων. Σταματώ εδώ, λέγοντας ότι σε κάποιες επιλογές και κάποιες προσαρμογές εξαρτώμεθα από τις ψηφοφορίες που θα γίνουν επί των άλλων εκθέσεων, που θα προηγηθούν και μετά από εκεί θα προκύψουν κάποιε τεχνικέ προσαρμογέ στο κείμενο και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι συμφωνίε που θα πρέπει να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Ξεκινά συζήτηση. Πολύ σημαντική αυτή η στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των συντονιστών. Ξεκινάμε του κοιόδης ηγητέ, ο σύθιστε George Lyon. έχει το λόγο, George. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Ζωβάνη Λαβία για τόσα μας είπε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Πάντως, η μέθοδος εργασίας είναι όπως και αυτή με τον ε, Καποσάντος που επικεντρωνόμαστε σε 4-5 άρθρα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ελπίζω να ακολουθήσουμε αυτή τη μεθοδολογία και για αυτό το θέμα. Έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες όσο γίνεται περισσότερο. Δεν έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες γιατί ο Τζοβάνι ευτυχώς έχει καθησυχάσει με το κείμενό του πολλές από τις ανησυχίες που είχα και ήθελα να υποβάλω με τροπολογίες. Οπότε με έχει καλύψει σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο ίδιος με τις δικές του τροπολογίες δηλαδή με κάλυψε. Θέλουμε ένα σύστημα που να βοηθάει για να έχουν καλή απόδοση και οι αγρότες και οι χώρες Με βέβαια ελέγχους, αποτελεσματικούς, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση των αγροτών στους κανόνες οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στις διαδικασίες έτσι όπως έχουν καθοριστεί αυτές και με ε, διαστευρωμένους ελέγχους επίσης. Θέλω να δω και τις κυρώσεις. Γιατί το θέμα δεν είναι αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει και δεν έχει υποβάλει ακριβώς όλα τα έγγραφα έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά κυρίως τι γίνεται με την χρηματοδότηση πώς τη Το θέμα της πολλαπλής ε, συμμόρφωσης πάντως δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις διαμαρτυρίες που ακούμε στις εκλογικές μας περιφέρειες. Γραφειοκρατία, δηλαδή ή άδικα πρόστιμα που επιβάλλονται. Αυτό ίσως μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι. Όντως, έχω και εγώ την αίσθηση ότι παρένε φορτωμένοι με γραφειοκρατία οι αγρότες και αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά στην κοινή γεωργική πολιτική. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον Τζοβάνι και τους άλλους σκιώδες θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Τζορτζ. Ο Λιντσέκ. Λουίς αντικαθιστά τον κύριο Έχεις το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να εξηγήσω γιατί ο κ. Σολενίτσακ ε, απουσιάζει. Είναι στην Επιτροπή Περιφερειακών ε, Θεμάτων και υποστηρίζει μια έκθεση της οποίας είναι ο εισηγητής. Θα έρθει οποια, όπου να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, μου ζήτησε να πω ορισμένα λόγια από τη δική του πλευρά. Προφανώς καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Λαδία για τον τρόπο με τον οποίο έχει συζητήσει με τους κοιοδησιητές. Έχουμε πολλά θέματα στα οποία υπάρχει μια σύγκληση και σύμνη απόφαση ε, απόψεων και πιστεύω θα συνεχιστεί αυτό. Επίσης, από την πλευρά της σοσιαλιστικής ομάδας εξακολουθούν να παραμένουν κάποια ερωτήματα, τα οποία ίσως θα πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευσης, ιδίως το θέμα των συστημάτων πληρωμής και των φορέων πληρωμής στον αγροτικό τομέα, και τα ερωτηματολόγια με τα οποία πρέπει να κάνουν αίτηση οι μικροί γεωργοί. Όλα αυτά είναι θέματα για τα οποία εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη διευκρίνηση των κειμένων που διέπουν τα θέματα αυτά και ιδίως θέλουμε να τονίσουμε το θέμα της απλοποίησης που είναι για μας ένα κομβικό θέμα. Τέλος, να πω ότι ο Τζοβάνι όταν είδε ότι πήρε μόνο 600 τροπολογία στην εκθεσή του δεν πρέπει να απογοητευτεί, δεν πρέπει να θεωρήσει ότι αυτό σημαίνει ίσονα σημασία της ε, εκθεσής του. Ίσα ίσα αυτό δείχνει την πολύ καλή ικανότητα του εισηγητή που αφαιρεί από τους συναδέλφους του την ανάγκη να καταθέσουν τροπολογίες και έχουμε κάθε διαθεσιμότητα να εργαστούμε μαζί σου Τζοβάνι για να μπορέσουμε να κλείσουμε και αυτό το θέμα στο γενικό πακέτο. Ευχαριστώ Λουίς. Συνεχίζουμε τους κοιόδης για τους πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την στάση του που είναι τόσο ανοιχτός. Όπως είπε και ο Τζόρτζ, ίσως να μην είναι το πιο ελκυστικό θέμα, αλλά είναι ένα από τα πιο σημαντικά στην μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γιατί εδώ συζητάμε κατά πόσο το δημόσιο χρήμα, μάλλον για το πού πρέπει να πηγαίνει το δημόσιο χρήμα. Υπάρχουν με εκλογικέ περιφέρειες βέβαια που θίγονται περισσότερο από άλλε, αλλά πάντως πάρα πολλέ όλε οι εκλογικέ περιφέρειες νομίζω ότι ανησυχούν για το πού πάει το δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα λοιπόν πρέπει να βγαίνει σε δημόσια αγαθά. Και αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μα ε, σε αυτήν την ε, έκθεση. Δεν πρέπει να γνωρούμε και μερικέ φορέ έχω την αίσθηση ότι το γνωρούμε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των δαπανών που πάνε στη Γεωργία και που δαπανώνται όμως εκτός Γεωργίας. Οι άνθρωποι μας παρακολουθούν τι κάνουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν με τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ έτσι ώστε το δημόσιο χρήμα να ε, δαπανάται αποτελεσματικά. Αλλιώς ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι πληρώνει για τα τρόφιμα, αλλά πληρώνονται οι αγρότες και από το δημόσιο χρήμα και μετά πρέπει να πληρώνουν οι καταναλωτές για ό,τι ε, προβλήματα κακής διαχείρισης έχουν προκύψει από τις πληρωμές που έχουν κάνει νωρίτερα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο πώς το σύστημα δουλεύει και πώς θα διασφαλίσουμε την δημοσιονομική αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους, όλες μας τις εκλογικές περιφέρειες, γιατί εμείς εκπροσωπούμε όλες και όχι μόνο μία. Να δούμε λίγο ότι επήγει αυτή, αυτή η κατάσταση. Αν δούμε λοιπόν τώρα τις προτάσεις της Επιτροπής και τις τροπολογίες που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο εισηγητής, έχω την αίσθηση ότι αν μιλάμε για τα συστήματα συμβουλών προς τους ε, γεωργούς, εδώ πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο με χρηστή διαχείριση. Γιατί τι έχουμε δει άλλο. Έχουμε δει ότι τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνονται για τη στρατηγική 2020, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για το 2020 είναι η χρηστή διαχείριση των κονδυλίων, η αποτελεσματικότητά τους. Άρα, σε όλες τις εξελίξεις που κάνουμε για την ΚΑΠ να έχουμε υπόψη μας την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και όταν συζητάμε για αυτά τα συστήματα ενημέρωση και συμβουλών προς τους αγρότες και εκείνα τα έχουμε υπόψη μας αυτό. Ενώ ο εισηγητής ασχολείται περισσότερο με τον ανταγωνισμό. Ενώ και η χρήση των φυσικών πόρων πρέπει εδώ να λαμβάνεται εξίσου υπόψη. Να πούμε ότι και αυτή η αποτελεσματικότητα είναι στοιχείο κλειδί. Τώρα για τις καλές περιβαλλοντικές ε, συνθήκες. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή κάποια πράγματα τα έχει βάλει στο πρασίνισμα. Το θέμα της εκπεριτροπής ε, καλλιέργειας κλπ. Αυτό αν σημαίνει ότι τελικά το πρασίνισμα δεν θα είναι πια υποχρεωτικό, αυτό σημαίνει ότι υποβάζουμε τις ε, προδιαγραφές μας. Γι' αυτό νομίζω εγώ ότι το πρασίνισμα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Και αυτό το τονίζουμε ξανά και ξανά. Έπειτα, το θέμα των ε, ειδών. Και εδώ είναι κάτι που το βγάζει ο εισηγητής. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι τα είδη που κινδυνεύουν από εξαφάνιση επηρεάζουν πάρα πολύ το οικοσύστημα. Είτε συζητάμε για πλημμύρε, είτε για ξηρασία, είτε για τέτοια. Αυτό παίζει ρόλο. Αν θέλουμε λοιπόν ένα καλύτερο ε, οικοσύστημα στο μέλλον, που να μην εξαρτάται από τα τεχνη, τεχνητά, ε, τις τεχνητές ε, ε, ουσίες λιπασμάτων, ε, πρέπει να φροντίσουμε τους φυσικούς πόρους. Αυτό που μας εκπλήσει επίσης είναι ότι ενώ προσθέτουμε εδώ την ε, οδηγία για το είδωρ και εκείνη για τα παρασιτοκτόνα, η Επιτροπή λέει ότι όλα αυτά πρέπει να λεφθούν υπόψη στην πολλαπλή συμμόρφωση μόνο εφόσον όλες οι χώρες έχουν καθορίσει προδιαγραφές που εφαρμόζονται στην Γεωργία. Δηλαδή, ενώ έχουμε συμφωνήσει πάνω σε κάποιους κανόνες για τη χρήση των παριστοκτώνων και για το είδωρ, βάζουμε τους αυτούς μας να εξαρτώνται από το πότε τελικά τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν για προδιαγραφές για τους αγρότες. Ελάθος! Η πολλαπλή συμμόρφωση υπάρχει εδώ γιατί όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβονται τον νόμο. Και οι οδηγίες αυτές εφαρμόζονται από το 2014, οπότε αποτελούν μέρος της πολλαπλής συμμόρφωσης. Τελεία και παύλα. Και εμάς μας εκπλήσει που τα βγάζει αυτά ο συγητή από την πολλαπλή συμμόρφωση λες και δεν παίζει πια κανένα ρόλο για τους γεωργούς ότι εμεί έχουμε ε, γκρίνει κάποιες οδηγίες. Όλοι πρέπει να τηρούν τον νόμο και οι αγρότες. Αλλιώς ο υπόλοιπο κόσμος θα μπορεί άλλη μια φορά για το τι κάνουμε με το δημόσιο χρήμα. Θέλουμε λοιπόν πιο εντατικές συζητήσεις πάνω σε αυτό και όχι να αρκεστείτε σε αυτό που είπαν οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές ότι θα συζητάμε ωραία και καλά και τι ωραία που τα καταφέρνουμε. Τώρα άλλα πράγματα που μας απασχολούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για παράδειγμα πάλι αυτό εξαιρέσει από την πολλαπλή συμμόρφωση. Εμεί οι πράσινοι πιστεύουμε ότι κανείς δεν πρέπει να εξαιρείται από την πολλαπλή συμμόρφωση. Κανένας. Όλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες και όλοι πρέπει να συμμορφώνονται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Συνεπώς δεν θέλουμε εξαιρέσει γι' αυτό. Για μας πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Ναι, κάποιοι λένε, α, ναι, και για τα βιολογικά προϊόντα. Ναι, και για τα βιολογικά προϊόντα. Εμείς είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτό. Όλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Τέλος, η πολλαπλή συμμόρφωση είναι κεντρικό θέμα για μας. Και δεν είναι κάτι που πλήττει την ΚΑΠ. Τώρα, οι συνάδελφοι από το ΕΛΚΑ, από την ΤΕΒΕ, σε γνωμοδότηση, η συγγήτρια εκεί είπε να μην πλήξουμε τις αρχές της κοινή γεωργικής. Μας έκανε εντύπωση που το ΕΛΚ, τουλάχιστον κάποιοι από το ΕΛΚ, βάζουν αυτό σε κεντρικό σημείο. Πολύ μας ικανοποίησε αυτό. Ελπίζουμε λοιπόν και εσείς να συμπεριλάβετε αυτή την αρχή, γιατί είναι και πολύ σημαντική για την πολλαπλή συμμόρφωση. Συνεπώς, όντως, την κυρία θα την πιέσουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να προχωρήσει πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Έπειτα, το πρασίνισμα ορισμένοι νομίζουν ότι είναι μόνο έξοδα. Ε, λοιπόν, όχι. Είναι για να αποφύγουμε ακριβώς το δημόσιο χρήμα που δαπανάμε δεν θα καταστρέφει την Ευρώπη, το περιβάλλον κτλ. Και να μην χρειάζεται να πληρώνουμε τρεις φορές μετά για να διορθώσουμε τη ζημιά που έχει γίνει από τον τρόπο με το οποίο καταρχήν δαπανήθηκε το δημόσιο χρήμα. Αυτή η αρχή λοιπόν είναι κεντρική σημασία και προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε με τις άλλες ομάδες αλλά και με ομάδες εκτός, αύριο για παράδειγμα, έξω από το Κοινοβούλιο που θα έχουμε μια πορεία για τα τρόφιμα και για το πώς δαπανώνται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Είναι αντίστροφα αναλόγω χρόνο αγόρευση με τη διάστηση της ομάδας των πρασίνων. Αυτό με ικανοποιεί τα μάλα. Καλό είναι να συλλέγουμε όλε τις ευαισθησίε. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μέγκελ, τον Γενικό Διευθυντή, και μετά θα ολοκληρώσει ο Τζοβάνι Λαβία. Α, και η Μαρία ζήτησε το λόγο. Η κυρία Μαγκίνα ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο μονάχα γιατί με ξύπνησε ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ξυπνήσατε και πάλι το ενδιαφέρον μου για το θέμα αυτό. Κάποια από τα σχόλιά σας δεν τα βρίσκω λανθασμένα, αλλά όλοι μας ανησυχούμε για τη δημόσια χρηματοδότηση. Αλλά και τα τρόφιμα είναι δημόσιο αγαθό. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι πολλές από τις πληρωμές προς τους γεωργούς είναι τμήμα του εισοδήματός τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν το κόστος παραγωγής έχει ανέβει ιδιαίτερα και αυτό είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην παραγωγή τρόφιμων. Αν εμείς μεταρρυθμίσουμε τη γενική αγροτική πολιτική με τρόπους που θα οδηγήσουν σε αύξηση της τιμή των τροφίμων, οι καταναλωτές σίγουρα θα αρχίσουν να χτυπάνε τις πόρτες μας. Εγώ λυπάμαι που δεν θα είμαι μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα διαπραγματευτούν αυτό το θέμα, και αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε τις απόψεις όλων. Σίγουρα είναι νόμος η πολλαπλή συμμόρφωση και κανείς δεν πρέπει να την χάνει ε, εξαίρεσης. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν θα εξαρτηθούν από το πώ θα πάει η συζήτηση για το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα. Αν οι γεωργοί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την οδό του πρασινίσματο, τότε τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλου στόχου. Α είμαστε λοιπόν πιο Προσεκτική για τα θέματα αυτά. Ακούσαμε πρόσφατα τα γεγονότα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί με, την, ε, με τις διάφορες ρυθμίσεις. Γραφειοκρατία πράσινη ή μη, όπως και να την αντιμετωπίσει κανείς. Έχουμε κανόνες οι οποίοι είναι ανθρώπινοι, είναι ανθρώπινη και εφαρμογή μπορούμε πάντα να τη βελτιώσουμε. Και σίγουρα δεν έχουμε αρκετά χρήματα στη διάθεσή μας για να καλύψουμε όλα τα προβλήματα. Όσο λοιπόν εξακολουθούν αυτές οι, οι διαφορές, μπορούμε πάντα να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας προς όφελος όλων των γεωργών και όλων των πολιτών στην Ευρώπη. Σήμερα το πρωί ήμουν σε ένα γεγονός όπου, σε μια εκδήλωση όπου αναφέρθηκε ότι παρά τις αυξανόμενες τιμές τροφίμων δεν μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερο να πληρώνουν περισσότερο οι καταναλωτές λόγω αυτής της γενικής κρίσης. Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή να είναι υπό απειλή και η χρηματοδότηση της γεωργίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τα προσθέσουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, οι γεωργοί έχουν προφανώς ένα πρόβλημα, αλλά και ο γενικός πληθυσμός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τα τρόφιμα. Σας τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε πόσο ευαίσθητα είναι όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να προστατέψουμε φυσικά και τα δημόσια χρήματα, τα δημόσια ταμεία. Ευχαριστώ Μάριαν. Ζητώ συγγνώμη από τον Ζαν Κάλο Σκοτά. Σε ξέχασα. Είσαι και ο Έχεις Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια που δεχτήκαμε τι εργασίε. Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Τα κάλυψε όλο και ο Σνταβία. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση για, το, για την πολιτική προσέγγιση και αυτά που λέει δείχνει ότι λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ζουν η αργιοργή μα. Γίνεται πιο εύληπτη για όλου του ενδιαφερόμενου στο τομέα εκείνη η αγροτική πολιτική. αρχή τη αναλογικότητα που συμπεριλαμβάνεται για το σύστημα επιβολή των κυρώσεων ακολουθεί την κατεύθυνση. Συμφωνώ και υποστηρίζω αυτή την πρόταση που απορρέει από το διάλογο το στενό που είχα και με τους γεωργούς στην περιοχή μου και εμεί σύμφωνοι. Και είναι κάτι που αντιστοιχεί με τι απόψει των γεωργών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδωσε συγκεκριμένε προτάσει ο συνάδελφο αντικατοπτεί στην πραγματικότητα εκατομμυρίων γεωργών που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που του επιβραδύνει στι δραστηριότητε. Για το πακέτο τη υπαίθρου είμαι και ω ηγητή και καλωσορίζω την πρόταση τη αυτόμα αποσύνδεση των ανάπτυξη υπαίθρου και μπορεί τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται από εκεί να χρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ Κάρλο. Δίνω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή τον κύριο Μέγκελ και μετά ο Τζοβάνι θα προβεί στην τελική του παρέμβαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να προσθέσω τις δικές μου ευχαριστίες στον κύριο Λαβία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση και έχει μια πολύ καλή βάση για την αντιμετώπιση των προτάσεων της Κομισιόν. Έχουμε πάντα Είχαμε πάντα την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά προηγουμένως με τον εισηγητή, να συζητήσουμε για όλα αυτά τα σημεία. Τώρα, ο οριζόντιος κανονισμός διαφέρει από, τους άλλους, από τις άλλες προτάσεις κανονισμού, γιατί καταρχήν είναι εγκάρσιος σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του αυτός ο κανονισμός και κατά δεύτερο λόγο έχει μεγάλη τεχνική πολυπλοκότητα. Ιδίω ό,τι αφορά τη, χρηματο, τη δημοσιονομική διαχείριση, τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για όσους πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κανονισμό. Γενικά, νομίζω ότι καλύπτει τρεις τομεί, είναι τρεις τομεί που θέλω να καλύψω μάλλον εγώ. Καταρχήν, Υπάρχουν προφανώς στοιχεία εξόχως πολιτικά σε αυτό τον κανονισμό και αυτό αντα... αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί. Αυτό αφορά την ε, ε, πολλαπλή συμμόρφωση, τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης, τα συστήματα κυρώσεων και το πρασίνισμα. Ένα δεύτερο σύμπλεγμα είναι τα ερώτηματα που αφορούν αυτούς που είναι περισσότερο τεχνικά μοιημένοι, αλλά έχουν και πολιτική σημασία σε σχέση με την δημοσιονομική διαχείριση, τον τομέα του λογιστικού ελέγχου, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Και μια τρίτη ομάδα είναι θεσμικά θέματα, πρόκειται για την εφαρμογή της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας, για τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Τώρα, ο οριζόντιος κανονισμός είναι μια ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την απλοποίηση της διαχείρισης της κοινή αγροτικής πολιτικής, τουλάχιστον να σκεφτούμε για το πώς θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό εμείς προσπαθήσαμε να παρέμβουμε και στις λεπτομέρειες του κανονισμού. Να απαντήσω και σε ορισμένα θέματα που αναφέρθηκαν, παραδείγματος χάρη το σύστημα διαβούλευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να έχει ένα σαφή χώρο εφαρμογή για να μπορέσει να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ε, διαβούλευση με τους ε, γεωργούς. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η διεύρυνση του συστήματος ή ο περιορισμός του συστήματος δεν θα ευνοήσει τη διατήρηση του, του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Επίσης για την πολλαπλή συμμόρφωση Υπάρχει φυσικά η υποχρέωση εφαρμογής για όλους τους γεωργούς. Τώρα, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, μια ισορροπία μεταξύ της απλοποίησης και της αποτελεσματικότητας, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε καλύτερα για τους γεωργούς οι οποίοι έχουν μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και το θέμα του αν θα πρέπει να τους επιβαρύνουμε με το σημαντικό άχθος της ε, πολλαπλής συμμόρφωσης, αυτό θα ακυρώσει κάθε μορφή της, ε, της απλοποίησης. Δεν πρόκειται για άρση της ανάγκης εφαρμογής της νομοθεσίας, απλώς τους, ε, θέλουμε να τους απελευθερώσουμε από το υπερβολικό άχθος γραφειοκρατίας. Ένα τρίτο σημείο σε σχέση με το θέμα αυτό, οι προτάσεις για την πολυετή διαχείριση Βλέπω στην αρχή να υπάρχουν απόψει οι οποίες είναι πολύ θετικές και σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ο πολιτή χαρακτήρα ήδη στους κανονισμούς μας γιατί η, οι γεωργοί ουσιαστικά μονάχα πρέπει να αντιμετωπίσουν μικρές διαφορές από το ένα χρόνο στον άλλο. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να μπορέσει αυτή η ιδέα να ενσωματωθεί περισσότερο στο κείμενο και να συμβάλλει στην επίτευξη της απλοποίησης. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο τομέα, τον τομέα που έχει να κάνει με τις τεχνικές ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να έχουν όμως επιπτώσεις στον πολιτικό τομέα. Πρόκειται για τα θέματα των ελέγχων που αναφερθήκανε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει και η αρχή της αναλογικότητας και να εφαρμόζεται πλήρως τα θέματα αυτά. Η αναλογικότητα αυτή εφαρμόζεται γέννη στα συστήματα κυρώσεων και πάλι πρέπει να δούμε πού μπορούν να προκύψουν περαιτέρω βελτιώσει. Αλλά θέλω να τονίσω ότι την ανάγκη διατήρηση ενό αποτελεσματικού καθεστώτο κυρώσεων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα κάνουμε βήματα προ το προς τα πίσω και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερα σφάλματα και περισσότερες ατασταλίες στο μέλλον. Ένα σημαντικό θέμα είναι οι κυρώσει που επιβάλλονται σε σχέση με το greening, το πρασίνισμα. Εδώ έχει προταθεί και νομίζω και ο εισηγητής το έχει ενσωματώσει αυτό, οι περιορισμοί, η, να υπάρξει περιορισμός των κυρώσεων μόνο για τον greening. <clears throat> Αλλά αυτό θα μας οδηγούσε σε μια κατάσταση όπου αυτή Συγγνώμη, να μην υπάρχουν κυρώσει για τον Green, πρότεινε ο εισηγητή, αλλά αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάσταση όπου αυτοί οι οποίοι δεν εφαρμόζουν το πρασίνημα δεν θα είχαν κυρώσει απλώς θα χάναν τα δυνητικά πλεονεκτήματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς για τον πολιτικό στόχο. Αν θέλει πραγματικά και το Κοινοβούλιο όπως η Κομισιόν να είναι υποχρεωτική η διαδικασία του πρασινίσματος, δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν κυρώσεις για τη μη εφαρμογή του. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η μείωση του διοικητικού άκτου και για τα κρατημέλη και για του γεωργού σε ό,τι αφορά του ελέγχους. Η πρότασή μα ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να μειώσουμε τους ε, ελέγχους εφόσον οι διοικήσει και τα συστήματα ελέγχου στα κρατημέλη λειτουργούν θετικά. Αυτό είναι σημαντικό και θετικό. Πρέπει όμω συγχρόνω να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ποσοτικούς ε, ενδείκτες που να καταδεικνύουν ότι τα συστήματα ελέγχου στα κράτη-μέλη λειτουργούν με σωστό τρόπο. Και να υπάρξει μια πρόταση η οποία θα εφαρμοστεί σωστά, ώστε να εξασφαλίσει ότι λειτουργεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, στο μέλλον θα πρέπει οι δηλώσει αξιοπιστία των κρατών μελών σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγροτικές, ε, οι αγροτικές ε, βοήθειες και επιδοτήσεις να έχει αξιόπιστο χαρακτήρα. Να έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε μια σωστή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη και να μπορούμε να έχουμε και εμπιστοσύνη στα στοιχεία τα οποία παρέχουν. Εάν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια σαφή σύνδεση και ελπίζω ότι και εσείς στην Επιτροπή σας το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, τότε μπορούμε στο μέλλον να μειώσουμε και να ε, ελαφρύνουμε τους ελέγχους για τους γεωργούς και τα κράτη-μέλη για το τρίτο σημείο που είναι η εφαρμογή των κανόνων της Λισαβόνας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει για το θέμα αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σαφώς θεσμικής και πολιτικής χρειάς. Εμείς παρακολουθούμε προσεκτικά αυτά τα οποία γίνονται σήμερα και βλέπουμε να υπάρχουν δύο αντίρροπες τάσεις οι οποίες αναδύονται. Ε, καταρχήν αυτά που η Κομισιόν θέλει ως εκτελεστικές εξουσίες να γίνονται όλο και περισσότερο <clears throat> κατεξουσιοδότηση πράξης και από την άλλη μεριά να αφαιρούνται δυνατότητες ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό είναι ένας δύσκολος τομέας. Δεν θέλουμε λοιπόν να επιλύσουμε αυτήν την ε, ε, συζήτηση σε ένα πρόωρο στάδιο γιατί δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τι συζητήσει οι οποίε θα εξακολουθήσουν σε πολιτικό επίπεδο για την ισορροπία μεταξύ πράξεων κατά και κατεκτέλεση. εκτέλεση. Τέλος, για το θέμα τη χρηματοδότηση αναφέρθηκαν τα 300 εκατομμύρια που, που θα μπορούσαν να επανεισαχθούν ω περιθώριο. Δεν έχουμε προτείνει ακόμα κάτι τέτοιο, γιατί αυτά τα 300 εκατομμύρια δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αντιμετώπιση εκ των περιστάσεων. Θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο αυτά τα χρήματα γιατί ε, θα πρέπει επίσης να σεβαστούμε την δημοσιονομική λιτότητα και να εξασφαλίσουμε ότι τα ποσά αυτά θα υπάρχουν αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ο εισηγητής αναφέρθηκε στο θέμα της εφαρμογής της αρχής νη συν 2 στα κατημέλη για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι θα αποσυνδέαμε με τον τρόπο αυτό τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, την εκτέλεση των προγραμμάτων και την χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Δεν μας φαίνεται αυτό ότι είναι μια θετική λύση. Έχουμε πάντα δυνατότητες να Έχουμε μεγαλύτερη ευκαμψία στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη και είμαστε πάντα έτοιμοι και εδώ μέσα στα πλαίσια του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να προτείνουμε λύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τελικό σημείο γενικό. Η πρόταση του 4% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγροτική ανάπτυξη αφορά οριζόντιες, ε, ε, είναι ένα οριζόντιο ποσό και υπάρχουν αυτές οι προτάσεις για 7% να φτάσει αυτό το ποσοστό στα 7% αλλά δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Και κλείνοντας να σας πω ότι πάντα είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε την τεχνική μας αρρωγή και εμπειρογνωμοσύνη και στο βαθμό του δυνατού να σας βοηθήσουμε στο έργο σας και να σας υποστηρίξουμε για την περαιτέρω επεξεργασία συμβιβαστικών τροπολογιών και ιδίως επειδή είναι ιδιαίτερα τεχνικό το θέμα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε εσά και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας εφόσον το επιθυμείτε για περαιτέρω συζητήσεις και περαιτέρω προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Γενική Διευθυντά Μέγκελ. Πολύ καλά έχουμε όλα τα στοιχεία. Τζοβάνι, αν θε ε, κλείσε με μια παρέμβαση σου και μετά πάμε στο τελευταίο σημείο τη μέση διάταξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιε χρήσιμε ενδείξει που απέρευσαν από τη συζήτηση. Σίγουρα τόνισαν, υπογράμμισαν κάποιε διαφορέ που υπάρχουν σαν αφορά προσεγγίσεις και μεταξύ πολιτικών ομάδων διότι κάποιος προσέχει πιο πολύ πραγματος χάρη την ανταγωνιστικότητα, άλλος τα περιβαλλοντικά, αλλά αυτό το γνωρίζαμε πριν ακόμα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να συγκεράσουμε αυτές τις θέσεις και δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Δύο ή τρία πράγματα θα ήθελα όμως να θίξω από αυτά που είπε στο τέλος ο Διευθυντής Μέκελ. Το θέμα του περιθωρίου όσον αφορά αυτό το περιθώριο δεν έχω τοποθέτηση σαν εισηγητής, δεν έχω τροπολογίες, είναι τοποθέτηση μιας πολιτικής ομάδας και νομίζω ότι δεν τη συμμερίζονται άλλοι σε αυτή την Επιτροπή. Ε, μάλλον τη συμμερίζονται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πιο περίπλοκο θέμα και που δεν καταφέραμε να επιλύσουμε όταν συζητήσαμε για την ευθυγράμμιση με τις συνθήκες της Αβώνας και παραμένει ε, ανοιχτό είναι το θέμα της ευθυγράμμισης. Ε, δεν έχω πρόβλημα να προβλέψω ποια θα είναι η θέση στο Κοινοβούλιο. Ήδη ψηφίσαμε, είχαμε μια θέση όταν είχαμε ψηφίσει την τοποθέτηση αφορά τον προηγούμενο οριζόντιο κανονισμό. Έναντι το συζητήσαμε με το Συμβούλιο είναι σημαντικό θέμα. Και αυτό αφορά τους κανονισμούς για αλλαγή της ΚΑΠ. Μπορεί να παραταθούν συζητήσει. Μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου βλέπουμε ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές. Και κάτι άλλο που δεν συζητήθηκε, αλλά είναι σημαντικό πιστεύω. Αυτό προσπάθησα να αναφέρω. Διάκριση μεταξύ απάτης και σφάλματος. Είναι μια σημαντική διαφορά, ουσιαστική. Χρειάζεται πιστεύω λοιπόν να εισαχθεί κάποιο εργαλείο, κάποιο μέσο, ένα σύστημα συναγερμού αν θέλετε, που να δίνει κάποια ένδειξη στο Γεωργό και λαμβάνοντα υπόψη την προσπάθεια απλούστευσης, αλλά να μην υπάρχουν και υπερβολικές κυρώσεις από την άλλη πλευρά έναντι των γεωργών που καμιά φορά μπορούν να κάνουν ε, κάποια μικρολάθη. Θέλω να συνεργαστώ βεβαίως με όλους τους εισηγητές, τους κοιόδης, για να φτάσουμε όλοι μαζί σε ένα κείμενο επί το οποίο συμφωνούμε όλοι. Πέρα από κάποια σημεία όπου υπάρχουν πιο βαθιές διαφορές, επί των άλλων, χωρίς δυσκολία πιστεύω ότι σύντομα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάληξη όσον αφορά τη συζήτηση και σε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστώ Τζοβάνι. Μετά μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για το πρωινό. Τα απόγευμα βεβαίως θα συνεχίσουμε στις 3 με τις διάφορες πρωτοβουλίες. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημείο 15 ενημέρωση από την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στις διεθνείς αγορές σιτηρών και τον αντίκτυπο στον τομέα της κτηνοτροφίας, ανταλλαγή απόψεων. Η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησε μια παρουσία πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αύξηση των τιμών στι αγορέ των σιτηρών και τι συνέπειε έχουν αυτέ οι αυξήσει στον τομέα τη κτηνοτροφία. Καλωσορίζω τον Διευθυντή Βεσλάινων τη Γενική Διευθύνσεω Άγκρι που θα μα συνοψίσει την κατάσταση και θα μα πει ποιε πρωτοβουλίε προτίθεται να δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Λοιπόν, να δώσω το λόγο καταρχάς το διευθυντή του κ. Σλάινερ και μετά ξεκινάμε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Στα μέσα ενημέρωσης ακούμε και διαβάζουμε ότι όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών, αν το συγκρίνουμε με την κατανάλωση, είμαστε αντιμέτωποι με ένα έλλειμμα το 2012-2013. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα που περιμένουμε για όλα τα σιτηρά παγκοσμίω στα τέλη της χρονιάς θα έχουν πέσει σε 380 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει 20% στην κατανάλωση. Άρα χάνουμε 1% στα από θέματα, δηλαδή από 20% σε 19% στα τέλη της χρονιάς. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία οδηγεί σε περισσότερες διακυμάνσεις στις τιμές. Κάτι το οποίο οφείλεται βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό στην ξηρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόεδρε, η κατάσταση εδώ είναι κάπως πιο ευνοϊκή από αυτή που υπάρχει παγκοσμίω ή στην Αμερική. Γιατί εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε μια συγκομιδή 279 εκατομμύρια τόνους. Κάτι το οποίο είναι 2% μόνο κάτω από το μέσο όρο για 5 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι μια λογική συγκομιδή. Συνεπώς, βέβαια ακόμα περιμένουμε την συγκομιδή για τον Αράσα ε, Αραβόστο λίγο παραπάνω, ε, για το ΣΥΤΟ επίσης περίπου στο μέσο όρο και για το κρυθάρι το ίδιο. Βέβαια, έτσι μπορούμε να έχουμε ακόμα ένα λεγόμενο πλεόνασμα εμπορίου 10 εκατομμυρίων τόνων. Συνήθως είναι 12-13 εκατομμύρια τόνοι, τώρα είναι 10 εκατομμύρια τόνοι. Έχει πέσει δηλαδή λίγο. Απόθεμα σημαίνει ότι εισάγουμε 13 εκατομμύρια και εξάγουμε 23 εκατομμύρια. Αυτό περιμένουμε για φέτος, γι' αυτό μιλάω για 10 εκατομμύρια πλεόνασμα κατά κάποιο τρόπο. Φυσικά έχουμε άμεση επαφή με την παγκόσμια αγορά. Οι εσωτερικές μας τιμές εξαρτώνται και από τις σχετικά υψηλές τιμές διεθνώς. Οι Ευρωπαίοι χρήστες σιτηρών εφαρμόζουν αντίστοιχες τιμές, όπως αυτές στην παγκόσμια αγορά. Πέρα από τα σιτηρά όμως υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τις πρωτεΐνες. Ε, σόγια, για παράδειγμα, στη συγκομιδή στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν χαμηλή. 670 δολάρια, ε, για παράδειγμα, για τη σόγια, που είναι η πιο σημαντική συγκομιδή πρωτεϊνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντως, περιμένουμε κάποια ανακούφιση σχετικά. Την άνοιξη του 2013, γιατί εξαιτία των υψηλών αυτών τιμών, Στη Νότια Αμερική δημιουργούνται διάφορες ε, μεγάλες ε, εκμεταλλεύσεις οι οποίες θα αρχίσουν ε, να αποδίδουν σύντομα. Τώρα για οποιαδήποτε άλλη παραγωγή, Πρόεδρε, αντιμετωπίζει σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής, γιατί βλέπετε ότι ένα μεγάλο μέρος των σύντρων που παράγουμε χρησιμοποιείται στις ζωοτροφές και η παραγωγή, η κτηνοτρόφη μάλλον, οι οποίοι βασίζονται σε τέτοιου είδους ε, ζωοτροφές, οι πρωτεΐνες, οι σιτρά κτλ, είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο. Έχουμε δει και κάποια αντίστοιχη κατάσταση. 2008-2009 είχαμε μια παρόμοια κατάσταση. Η διαφορά όμως με τότε όσον αφορά την κτηνοτροφία είναι ότι σήμερα οι τιμές για τα ζωικά προϊόντα είναι σχετικά υψηλές, κυρίως για το κρέας. Αν δείτε τις τιμές για τα βοηδή, για το βόηο κρέας, 4.000 ευρώ το τόνο περίπου. 180% της τιμής παρέμβασης. Οι τιμές του χείρου κρέατος επίσης είναι υψηλές και των πουλερικών. Βέβαια είναι και συγκυριακό. Είδατε ότι είχαμε την απαγόρευση της παραγωγής εκλοβούς ε, στοιχείες κλοβών όσον αφορά τα πουλερικά, κάτι το οποίο οδήγησε επίσης σε υψηλές τιμές. Και όσον αφορά το χείριο και το βόλιο, οι τιμές αυτές έχουν να κάνουν και με τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Συγκυριακά συνεπώς μιλώντας, οι τιμές είναι υψηλές και η παραγωγή μας άρα έχουν λίγο παραπάνω δυνατότητες θα έλεγα να απορροφήσουν αυτές τις ε, ψηλές τιμές των καταναλωτή. Όμως Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις ζωοτροφές ε, βλέπουν τις τιμές ε, μάλλον να μειώνονται. Για το κρέας πάντα, ε, για το γάλα τώρα. Οι τιμές έπεσαν παγκοσμίω μετά από δύο χρόνια ιδιαίτερα υψηλές τιμές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είχαμε παραγωγή περισσότερου γάλακτος εξαιτίας των υψηλών τιμών, οπότε χρειάστηκε να απορροφηθεί το επιπλέον γάλα, κάτι το οποίο επέδρασε στις τιμές. Οι τιμές πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν έπεσαν κάτω από το 120% του επίπεδου ασφαλείας. Το 2008-2009 ήμασταν περίπου σε αυτό το επίπεδο, αλλά πριν τις θερινές διακοπές ήμασταν στο 120% και παραπάνω για τη σκόνη γάλακτος για παράδειγμα. Από τον Ιούλιο οι τιμές αυξάνονται για το γάλα. Είναι και εποχιακό, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι οι τιμές παραγωγής αυξάνουν. Πάντα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις αυξήσεις αυτές ε, το, η παραγωγή γάλακτος και τις τιμές γάλακτος που πληρώνουν οι καταναλωτοί, αλλά οι τιμές τώρα πάνε στο 31 σεντ κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τιμές Ιουνίου-Ιουλίου. Τιμές που βλέπουμε στις αγορές που μας λένε περισσότερα για τις τάσεις εκεί βλέπουμε αυξήσεις. Το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, στην Ιταλία είχαμε μια αύξηση 19%, Βόρεια Ιρλανδία 21% και στις κάτω χώρες 64%. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια αύξηση στην τιμή του γάλακτος. Κάτι άλλο που απορρέει από την ξηρασία στις ΗΠΑ είναι ότι η παραγωγή γάλακτος μειώνεται στις ΗΠΑ που σημαίνει ότι οι δικές μας εξαγωγές έχουν περισσότερα περιθώρια σε αυτή την αγορά, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί τότε θα μπουν στο παιχνίδι και οι φίλοι μας από τη Νέα Ζηλανδία. Συνεπώς είμαστε αισιόδοξοι ότι οι τιμές αυτές που έχουν να κάνουν και με τις καλές επιδόσεις μας στις εξαγωγές θα συνεχιστούν σε θετική τάση. Τέλος, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα σιτηρά, η κατάσταση είναι κάπως δύσκολη. Υπάρχει κίνδυνος ε, για τις τιμές εξαιτία ε, των χαμηλών αποθεμάτων, κάτι που δημιουργεί αστάθεια. Η κατάσταση τώρα για τους αγρότες εξαρτάται από το σε τι βαθμό εξαρτώνται από τις ε, ζωοτροφές. Και η κατάσταση διαφορετική στον Νότο και στο Βορρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως προσπαθεί να συνεισφέρει και να ανακουφίσει κάπως ε, την κατάσταση. Διεθνώς ε, διαπιστώνουμε ότι και παγκοσμίω οι τιμές είναι όπως αυτές που έχουμε και εμείς. Θέλουμε λοιπόν διαφάνεια και είναι προσπάθειες που κάνουμε ε, συνεχώς για να αποφεύγεται περιττή κερδοσκοπία βάσει του τι υπάρχει ως απόθεμα και τι δεν υπάρχει. Γι' αυτό θέλουμε τη διαφάνεια. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει ιδιαίτερα θετικό ρόλο για να ε, διασφαλίσει ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα αποθέματα σιτηρών. Όσον αφορά τις εισαγωγές μας τώρα, τους δασμούς τους εισαγωγικούς. Βάζουμε 0, μηδενικό επίπεδο, και βάσει του υπολογισμού που κάνουμε για τον αραβόσιτο, ακόμα και εκτός ποσοστώσεων, για τον αραβόσιτο είναι μηδέν. Άρα το περιθώριο για εισαγωγές ζωοτροφών, μεγάλες ε, εισαγωγές είναι ανοιχτό. Ελέγχουμε βέβαια την κατάσταση και ίσως στις αρχές της επόμενης χρονιάς να πάρουμε επιπλέον μέτρα για να υπάρξει δυνατότητα και άλλων εισαγωγών σιτηρών για ζωοτροφές. Αυτά προς το παρόν. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε και που μας παρουσιάσατε αυτές τις πληροφορίες. Άλλος της αγορεύει βούλετε. Ερωτήσεις. Ορίστε. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Μόνο ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς την Κομισιόν. Είχατε κάνει μια ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Κομισιόν θα αλλάξει τα σχέδιά της σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα. Η, από την στρατηγική να καλύψουν 10% τα βιοκαύσιμα φαίνεται ότι η Κομισιόν σκέφτεται να, μετα... να τροποποιήσει αυτή την ε, αλλαγή. Δεν έχετε αναφέρει όμως τίποτα για το θέμα αυτό. Και αυτό το θέμα των βιοκαυσίμων έχει επιπτώσεις στις, ε, στις αγορές ή δεν έχει κάποια επίπτωση. Τι, τι, θέλετε λοιπόν να κάνετε. Θα μειώσετε το στόχο του 10% στα 5% ως στόχο για τα βιοκαύσιμα. Επίσης για τον τομέα γάλακτος είπατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν, έχει επίσης φτάσει, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο του δικτύου ασφαλείας. Αλλά ε, λέτε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός ε, ε, ανάγκης στα 20 cent. Είναι αυτό ακριβές ή θα γίνει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Κάποιο άλλο θα ήθελε να λάβει το λόγο, να θέσει κάποιο ερώτημα. Όχι. Δίνω το λόγο λοιπόν και πάλι στον εκπρόσωπο της Επιτροπής για να απαντήσει στο σαφές αυτό ερώτημα. Παρακαλώ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ καιρό. μικροφώνου Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν γνωρίζω αν υπήρξε αλλαγή όσον αφορά τους στόχους που αποφασίστηκαν για τα βιοκάψιμα μέχρι το 2020. Φαντάζομαι ότι διεξάγονται συζητήσεις από αυτού. Απ' την άλλη θα έλεγα ότι βέβαια οι τιμές της αγοράς θα καθορίσουν σε το βαθμό ε, στον οποίο θα απορροφούνται και τα ζητούνται τα βιοκαύσιμα. Αν θέλει κανείς να παράγει ενέργεια βάσει των ακριβών σιτηρών, θα κοστίζει ενέργεια. Και πρέπει να αποφασίσει η αγορά προς τα που θα κινηθούν τα σιτηρά. Συμφωνώ με τον κύριο Χάουσλινγκ όμως ότι αυτή η πολιτική μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των σιτηρών. Και στη ΣΥΠΑ έχει συνέπειες όπου υπάρχουν σημαντικότερα προγράμματα όσον αφορά τον αραβόσιτο για να χρησιμοποιείται για βιοκαύσιμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση των σιτηρών στα βιοκαύσι... η χρήση των βιοκαυσίμων σχετικά μικρή, υπάρχει επιρροή, αλλά είναι μικρή. Όσον αφορά το γάλα, ναι, πράγματι, το κόστος για τον παραγωγό αυξάνεται κυρίως για εκείνους που βασίζονται σε ζωοτροφές που αγοράζονται απ' έξω από την εκμετάλλευση, εξαρτάται και από την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, όλη, αυτή η εξίσωση. Όπως είπε και ο Σέστριγκερ, η τιμή του δικτύου ασφαλείας είναι 21,5 cents και η τιμή αγοράς είναι περίπου 13 cents. Άρα είναι 10 cents πάνω από το δίχτυ ασφαλείας. Αν δείτε τα διάφορα εργαλεία για την αγορά που έχουμε στην διάθεσή μας όπως ιδιωτική αποθεματοποίηση σε παρέμβαση Είχε ανοίξει μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου, αλλά ήταν πιο ψηλέ οι τιμές από τις τιμέ παρέμβαση, άρα δεν προσφέρθηκε κανείς για παρέμβαση. Λογικότατο αυτό. Δεν χρειάστηκε η χρήση του εργαλείου αυτού. Όσον αφορά την αποθήκευση του βούτυρου, χρησιμοποιήθηκε το μέτρο αυτό για 100.000 περίπου τόνους που ξαναγοράζονται και διατίθεται στην αγορά τώρα. Τα διάφορα διθέσιμα μέσα λοιπόν λειτουργήσαν. Εξαγωγικές επιδοτήσεις με τόσο ψηλές τιμές είναι καταρχήν διαθέσιμες, δεν τις ζητά κανείς όμως. Διότι η διαφορά με τις τιμές παγκόσμιας αγοράς δεν δικαιολογεί εξαγωγικές επιστροφές. Για την ώρα η αγορά πρέπει να βρει τη δική της ισορροπία στον τομέα των γαλακτοκομικών. Όταν είσαι πάνω από 130% του επίπεδου του δικτύου ασφαλείας, ε, δεν μπορεί να πεις ότι περνάς κρίση. Είσαι σε μια κατάσταση όπου οι τιμές είναι σχετικά ψηλές. Δεν αρνούμε ότι οι τιμές των ζωοτροφών είναι επίσης υψηλές, οπότε μειώνονται τα περιθώρια. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Δεν υπάρχουν ας ερωτήσεις από τους συναδέλφους, άρα μπορούμε τώρα να διακόψουμε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση από αυτού του σημείου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας παρουσιάσει υπομορφή ενός σημειώματος, υπομορφή εγγράφου εργασίας που θα δώσει στη γραμματεία κάποιες πληροφορίες, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουν και άλλοι συνάδελφοι τις πληροφορίες. Αναφέρομαι σε έγγραφα εργασία, σημείωμα εργασία, διότι οι πληροφορίε που μας δόθηκαν ήταν προφορικέ τώρα. Ξανασυναντιόμαστε στις 3, εδώ. Ο κύριος Αλετράρης, ο Κύπριος Υπουργός, θα είναι παρόν. Και στις τρεις και μισή θα συνεδριάσουν οι συντονιστές μέχρι τις 4 και 30, 3 με 4 και 30. Οι εκπρόσωποι των επιτροπών που γνωμοδοτούν επί της εκθέσεώς μας θα συναντηθούν εδώ και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.